Liebe Kollegen, liebe πολυάριθμοι συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε ίσως. Δεν... είναι εδώ ακόμη ο οπότε ίσως θα μπορούσαμε να αλλάξουμε ίσως τη σειρά. Μπορούμε να περάσουμε στο θέμα 2. Καλή ιδέα είναι αυτή που Ίσως είναι η μόνη μέθοδος την οποία θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε. Βλέπω τον εισηγητή του σημείο 15. Δεν ξέρω όμως αν είναι ισχυώδης εδώ παρόντες. einen Vorschlag machen. Äh, Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με το σημείο 15. Η έκθεση του κ. Μανκεβιτς. Γιατί ή αποτελεί κάποιο πρόβλημα για τους άλλους συναδέλφους. Γίνεται. Ωραία, μπορούμε να αλλάξουμε τότε τη σειρά. αλλά λείπουν πολλοί συνάδελφοι δυστυχώς Μπάλιαν βάζει και μετά θα ενοχληθούν που το θέτω πρώτο σημείο στη μέση διάταξη και θα είναι παρόντες. I think is not going to be here δεν θα έρθει και αυτή. Πάμε, ξεκινάμε. Ξεκινάμε το σημείο 13. Η έκθεση Έτλερ. Ίσως πρέπει να πάμε λίγο πιο γρήγορα. Έχουμε τρία σημεία στη μέση διάταξη πριν από την ε, ψηφοφορία και πρέπει να είναι κάπως σύντομη η συζήτηση. Κρίστιαν, στα γρήγορα, στα γρήγορα. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, εφόσον χθε ήσασταν γενναιόδωρο μαζί μου που ήμουν σκιώδη εισηγητή, τώρα θα προσπαθήσω να είμαι πιο σύντομο σαν εισηγητή. Βλέπω ότι δεν υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θα έχουν να προσφέρουν στη συζήτηση. Και εξάλλου ήταν πολύ καλή η συνεργασία μας με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ αλλά η Επιτροπή μας, η Επιτροπή Βιομηχανίας δεν έχει τόσο πολύ εμπλακεί στο θέμα αυτό γιατί εξακολουθούν να παραμένουν ορισμένα νομικά θέματα Εγώ θα ήθελα λοιπόν να μιλήσετε με την κυρία Χολμάιερ και να της πείτε ότι θα πρέπει να εμπλακεί λίγο περισσότερο η Επιτροπή Βιομηχανίας, η Ήτρε, ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε και ένα πλαίσιο ολοκληρωμένο για την αντιμετώπιση του κυβερνού εγκλήματο και να κλείσουμε όλα τα παραθυράκια και τι κερκόπορτέ. Έχουμε αντιμετωπίσει μια σειρά προβλήματα. το <clears throat> λεγόμενο πρόβλημα track and trace, η ανείχνευση δηλαδή της προέλευση μια ε, απειλής ή μιας ε, κυβερνοεπίθεσης. Αυτό όμω είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο στην πραγματικότητα. Και επομένως ε, η έκθεση της κυρίας Χολμάιερ είναι, ακόμα και αν είναι σε εμβριακή ακόμα μορφή, μια πάρα πολύ σημαντική έκθεση για την αντιμετώπιση της ε, κυβερνο της κυβερνοεγκληματικότητας η οποία έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην Ευρώπη, ζημίες δισεκατομμύριων ευρώ, περιπτώσεις που έχουν έρθει ενώπιον των δικαστηρίων κτλ. Εμείς στην γνωμοδότηση ε, επομένως διεκδικούμε μια σωστή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση για τα θέματα αυτά. Αναφέρομαι τα οικονομικά προβλήματα, του οικονομικού κινδύνους που μπορεί να επέχει η κυβερνοεκκληματικότητα για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, και οι οποίε από μόνε τους δεν έχουν την οικονομική επιφάνεια για να προβούν σε μέτρα προστασία. Επίση, τονίζουμε τη διεθνή διάσταση του προβλήματο στην ανάγκη να υπάρξει συνεργασία και συντονισμό με άλλε χώρε και άλλου οικονομικού ομίλου. Και επομένω είναι απαραίτητο να υπάρξει και μια γενικότερη αντιμετώπιση για τα θέματα αυτά ε, η χρησιμοποίηση βέβαια στοιχείων από το ίντερνετ γίνεται και από εταιρείε οι οποίε δεν έχουν εγκληματικού στόχου, το κάνουν για διαφημιστικού ή άλλου λόγου προβολή. Θα πρέπει να κάνουμε την απαραίτητη διαφοροποίηση μεταξύ αυτών και των εγκληματικών οργανώσεων και να του επιτρέψουμε να έχουν ένα πλαίσιο λειτουργία. Ευχαριστώ. Κύριο Ένσο, έχει το λόγο. Ε, Σας ευχαριστώ και εγώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να χαιρετήσω τη γνωμοδότηση του κυρίου Έλεα και να τον ευχαριστήσω για την εργασία του μέχρι τώρα. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πακέτο νομοθετικού χαρακτήρα σε ό,τι αφορά την αποτροπή κυβερνοεπιθέσεων και πιστεύω ότι η γνωμοδότηση του κυρίου Έλερ αντιμετωπίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα σημεία τα οποία και εμείς θα θεωρούσαμε πιο σημαντικά στον τομέα αυτό και είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε <clears throat> την γνωμοδότηση στα γενικά της στοιχεία. Όπως είπαμε και χθε. Όπως είπαμε και χθε σε σχέση με την ΕΝΗΣΑ, είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει σωστή κατανομή αρμοδιοτήτων και η ΕΝΗΣΑ να συνεχίσει να έχει ένα σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των ε, κυβερνοεπιθέσεων αυτών γιατί ο εντοπισμός των κινδύνων μπορεί να είναι σχετικά απλός, αλλά αυτό από μόνο του δεν αποτελεί ένα προπήριο, ένα φράγμα στις επιθέσεις αυτές. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τον κύριο Έλερ. Άλλοι θέλουν να λάβουν το λόγο, δεν βλέπω κανένα. Η κυρία Μαντουρέλ. Μαντουρέλ. Eh, Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα μόνο να θυμίσω κύριε Πρόεδρε ότι είναι ουσιαστικότατη αυτή η οδηγία για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στις Βρυξέλλες ε, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε την καλύτερη λειτουργία των ε, σύστηματων πληροφοριών. Είναι ουσιαστική αυτή η υποστήριξη της κοινωνίας της πληροφόρησης για να προωθήσουμε την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη. Όπως είπε όμως ο προλαλής σας, ο αγώνας κατά των ε, πληροφορικών επιθέσεων είναι μόνο ένα τμήμα της γενικότερης στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εγγυθεί την ασφάλεια των ε, συστημάτων επικοινωνίας και πληροφόρησης. Εδώ έχουμε και άλλα ρίσκα, τη δυσλειτουργία για φυσικά φαινόμενα ή για ανθρώπινα λάθη. Βέβαια τα προβλήματα τεχνικής, ε, ε, τα προβλήματα πληροφορικής ξεπερνούν τα σύνορα θα πρέπει λοιπόν να προσεγγιστούν, να προσεγγιστούν μεταξύ τους τα ποινικά συστήματα των κρατών μελών, να βελτιώσουμε την δικαστική συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών. Εγώ κύριε Πρόεδρε είμαι η εισηγήτρια στην, στην ΣΕΝΤΕ εκ μέρους της ομάδας μου για αυτό το θέμα και θα σας παρουσιάσω εδώ σύντομα μερικές από τις τροπολογίες που θα παρουσιάσω στην ΣΕΝΤΕ και που έχουν ως στόχο να εξάρουν τη σημασία των τεχνολογιών πληροφόρησης και πληροφορικής και το ρόλο που παίζουν για την ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών και για τις επιχειρήσεις μας. Επίσης θέλω να τονίσω ότι η απειλή ε, επιθέσεων στα συστήματα πληροφορικής είναι μια πραγματική απειλή πολύ σοβαρή που χρειάζεται συντονισμένη απάντηση από την Ευρώπη. και η σωστή τους ε, λειτουργία αποτελεί πυλώνα της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Έλεγα πριν ότι οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και πληροφόρησης ξεπερνάνε τα εθνικά μας σύνορα. Χρειάζεται συντονισμός, έχουμε όμως και τις απειλές διεθνών επιθέσεων, θα πρέπει η Ευρώπη να εντείνει τη διεθνή συνεργασία, πρόκειται για οικουμενικά προβλήματα που χρειάζονται οι οικουμενικές λύσεις ο συντονιστής για την κυβερνητική κυβερνοασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Και θα πρέπει να υποστηριχθεί. Ο, κύριος Μπιτικόφερ. Για να επιταχύνω τη διαδικασία, λέει ο κύριος Μπιτικόφερ. Ε, δεν χρειάζομαι να λάβω το λόγο. Για να επιταχύνω τη διαδικασία θέλω να σας εξοικονομήσω χρόνο αγόρευσης και δεν θα λάβω το λόγο. Ωραία. Αυτό είναι πολύ καλό. Άλλες ε, παρατηρήσεις, άλλες, άλλες παρεμβάσεις. Ο κύριος Έλερ θέλει να πει κάτι τίποτα. Η Κομισιόν ούτε και αυτή. Πάει αυτό το σημείο λοιπόν της ημερησίας διάταξης. Πάμε στο σημείο 14 κατά συνέπεια. Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα εμπορική ισορροπία. Στις 11 Οκτωβρίου, στις 12 η ώρα, είναι η προθεσμία κατάσταση τροπολογιών για την έκθεση ΕΛΕΡ. 14 λοιπόν, η ισορροπία, η έλλειψη ισορροπίας. Ο κύριος Ζαντό είναι ο μόνιμος εισηγητής μας, είναι παρόν, έχει και το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, καλημέρα σε όλους. Για αυτήν την έκθεση δεν έχουμε ακόμη την έκθεση πρωτοβουλία στη σύντα της κυρίας Δεσαρνές, όμως ορισμένα αρχικά σημεία. Πρώτον, η τεράστια ανισορροπία των εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. Ανισορροπία που έχει αρχίσει και τονίζεται κυρίως στον τομέα των εμπορευμάτων η Ευρώπη είναι καθαρή εξαγωγέας ως επενδυτής, αλλά στο εμπόριο, στην ανταλλαγή των εμπορευμάτων έχουμε τεράστια προβλήματα. Προβλήματα τα οποία συνδέονται κατά τη γνώμη μας με, πολλές, με πολλές ε, πτυχές οι οποίες έχουν να κάνουν και με θεσμικά προβλήματα. Η Ευρώπη μη έχοντας μία σαφή βιομηχανική πολιτική. Η Ευρώπη η οποία δρά διαιρεμένη έναντι της Κίνας, το βλέπουμε εξάλλου κάθε φορά που έχουμε επισκέψεις της κινέζικης κυβέρνησης, κάθε αρχηγός κράτους ή κυβέρνηση στην Ευρώπη, είναι πάντοτε πανευτυχής να υπογράφει μερικά συμβόλαια, υπερτιμημένα πολλές φορές ως προς αλλά δεν υπάρχει μια συνολική προσέγγιση των Ευρωπαίων έναντι της Κίνας η Κίνα μας διαιρεί πολλές φορές σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ακριβώς λόγω της έλλειψης βιομηχανικής, πολιτικής και συντονισμένης προσέγγισης έναντι, έναντι της Κίνας δεν μπορούμε να απαντήσουμε στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που μας θέτει η Κίνα. Εμείς σε αυτήν την γνωμοδότηση τονίζουμε μερικά πράγματα. Ένα, αυτήν την πρόκληση για συντονισμό που δεν μπορεί παρά να βασιστεί σε μια ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική η οποία είναι πάντοτε απούσα. Δεύτερο, ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που οφείλεται στη διαφορά του οικονομικού και κοινωνικού μοντέλου της προστασίας των μισθωτών προστασία της ε, πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτό είναι και το πιο γνωστό πρόβλημα. Και σήμερα αυτό το θέμα βρίσκεται στο επίκεντρο συζήτηση στην ε, Επιτροπή, στην Επιτροπή Απασχόλησης. Επίσης τα κλήρων. Η, η έλλειψη των κληρονομικών ε, κληρονομικού δικαίου στην Κίνα δημιουργεί προβλήματα και τέλος πάντων ε, οδηγεί σε μία στάση ε, που από τη δική μας τη μεριά μια στάση πολλές φορές προστατευτική. Θα πρέπει εμείς να θέσουμε τους όρους μας για την πνευματική ιδιοκτησία, για τους υγειονομικούς κανόνες, για τους κοινωνικούς κανόνες και να δώσουμε μια άμεση βιομηχανική απάντηση με, την, με μια βιομηχανική ευρωπαϊκή πολιτική και η Ευρώπη να σκεφτεί με σε έναν τρόπο ερεσιμότητας των ανταλλαγών με την Κίνα σε περίπτωση που οι ανταλλαγές αυτές δεν ανταποκρίνονται ε, στις, ε, στα ζητούμενα που πρέπει να γίνονται σεβαστά για θέματα ε, περιβαλλοντικά, για θέματα κλίματος, για θέματα κοινωνικά, για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Ευρώπη και η Κίνα είναι δύο ήπειροι, λέει ο μιλητής, ε, πολύ φτωχές ε, φυσικούς ε, πόρους για τις προκλήσεις της πράσινης οικονομίας, της τεχνολογίας. Έχουμε την δυνατότητα καταπληκτικών εταιρικών σχέσεων όταν είμαστε διασφαλισμένοι στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας για τη μεταφορά τεχνολογίας. τότε μπορούμε να προτείνουμε μια πραγματική εταιρική σχέση με την Κίνα. Πρόκειται λοιπόν για μια διάγνωση αρκετά κακή ε, για την ικανότητα της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης να διαπραγματευτεί με την Κίνα, έλλειψη συντονισμού, έλλειψη σαφούς βιομηχανικής πολιτικής, έλλειψη συστημάτων προστασίας ε, των ε, μισθωτών τόσο στην Ευρώπη, στην Κίνα, ε, η υγειονομική προστασία, προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Και από την άλλη μεριά διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις σύναψης εταιρικών σχέσεων γύρω από την πράσινη οικονομία και την τεχνολογία που θα μπορούσαμε να αναλάβουμε από κοινού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Πυρίλο. Συγγνώμη, συγγνώμη που καθυστέρησα. Ξέρω ότι πρόκειται για μία εκπληκτική έκθεση. Σημερίζομαι όλη την ε, οπτική και όλα τα σημεία. Η Κίνα είναι ένα σημαντικός ε, οικονομικός και εμπορικός εταίρος για την Ευρώπη και οι σχέσεις σίγουρα πρέπει να ενισχυθούν, αλλά υπάρχουν ακόμη μερικές πλευρές ε, που μας εμποδίζουν στη σύναψη εμπορικών σχέσεων με, βασισμένες στην αρχή της αμοιβαιότητας. Για το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας. Παρά τις σημαντικές πρόοδους της κινέζικης νομοθεσίας, παραμένει ακόμη προβληματική εφαρμογή τους. Εγώ εύχομαι η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνα, που ε, στοιχίζει 16 ε, ευρώ, 16 εκατομμύρια συγγνώμη ευρώ να αποτελέσει το πρώτο βήμα στη συνεργασία. και θα μας επιτρέψει να έχουμε προϊόντα στην αγορά στη σωστή τιμή. Να. Η τιμή να περιλαμβάνει και το ερευνητικό κόστος και το κόστος κατασκευής ε, των προϊόντων μας. Έχουμε επίσης ε, τους ειδικού ε, δασμούς για τις πρώτες ύλες όπως επίσης και την περιορισμένη δυνατότητα του να συμμετέχουν ξένες επιχειρήσεις σε διαγωνισμούς και δημοπρασίες στην Κίνα. Πολλοί κλάδοι της ε, κινέζικης οικονομίας ε, είναι απαγορευμένοι για τις ξένες επιχειρήσεις. Η Κίνα κάνει ό,τι μπορεί για να ε, μη σέβεται, για να μην σεβαστεί τη μεταφορά τεχνολογίας και know-how, την αμοιβαιότητα αυτής της μεταφοράς. Υποστηρίζω ότι για κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα θα πρέπει να εφαρμόσουμε νέες διαδικασίες μεταρρύθμισης, για να έχουμε δηλαδή αηφόρες διαδικασίες και θα παρουσιάσω κατά συνέπεια τροπολογία στην έκθεση. Ευχαριστώ πολύ κύριο Χόλ. Κύριε Χόλ συγκεκριμένα. Καλωσορίζω αυτήν την έκθεση και συμφωνώ με τα σχόλια που ακούστηκαν. Βέβαια, πράγματι υπάρχει λόγος να ανησυχούμε για κάποιες από τις προστατευτικές πολιτικές ε, που εφαρμόζει η Κίνα. Εγώ θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για κάποια σημεία, όπω είναι ο τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε πιθανά να αντιμετωπίσουμε πόρου όπως οι σπάνιε γέε και πώ μπορούμε και εμεί να βελτιώσουμε τη συνολική μα στρατηγική και την ανακύκλωση και τη χρήση αυτών των νέων πόρων. Πολλά μπορούμε να κάνουμε για να ξεπεράσουμε το πρόβλημα των κινέζικων περιορισμών στο θέμα αυτό. Έχω όμως μια ανησυχία σε σχέση με την παράγραφο 3 συγκεκριμένα. Νομίζω ότι στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά είμαστε οι ευεργέτες στις εμπορικές σχέσεις. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες απέναντι στην Κίνα. Δεν θα πρέπει να ακολουθήσουμε κι εμείς ε, το μονοπάτι του προστατευτισμού Καταλαβαίνω το πρόβλημα που υπάρχει με τα αγαθά τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά που ουσιαστικά ε, δεν ε, συμφωνεί η συσκευασία τους με αυτά τα οποία πραγματικά κάνουν. Στην παράγραφο 3 συγκεκριμένα ε, που ζητεί τη σταδιακή εισαγωγή επιβολή όρων ή προσαρμογή στα σύνορα ω προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα δεν με βρίσκει σύμφωνη. Θα έπρεπε νομίζω αντίθετα να επικεντρωθούμε στην ε, επιτήρηση, στην εποπτεία τη ε, δική μα αγορά. Σίγουρα υπάρχουν παράπονα από του κλάδου, από τη βιομηχανία οι πρόσωποι της λένε ότι δεν γίνονται αρκετά πράγματα ώστε τα προϊόντα που κυκλοφορούν, που εισάγονται στην αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σίγουρα αν συμμορφώνονται ή όχι προς τα κοινοτικά πρότυπα όπως θα έπρεπε. Μια από τις δυσκολίες είναι ότι η επιτήρηση, η της αγοράς είναι εθνική αρμοδιότητα και είναι δύσκολο να εξασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη-μέλη θα διαθέσουν τους απαιτούμενους πόρους ε, στα ε, αρμόδια γραφεία. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε αρκετά προσεκτικά πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την εποπτεία των αγορών και να δούμε κατά πόσο μπορούμε να κάνουμε κάτι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε κάθε κράτος μέλος, οποιοδήποτε ε, κράτος μέλος, θέλει να συνεργάζεται και να ε, έχει συναλλαγές εμπορικές με την Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να τηρεί και να συμμορφώνεται προς κάποια πρότυπα και να υπάρχει ισότιμη εμπορική σχέση όπως και με την Κίνα βέβαια στην προκειμένη περίπτωση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καιρός είναι πια. Καιρός πια είναι να έχουμε μια τέτοια έκθεση και αυτό το είπε και στη χώρα μας δηλαδή ένας κομμουνιστής καθοδηγητής στη 1.900 δις δολάρια διέθετε στα αποθέματά της η Κίνα πριν από χρόνια και έλεγε ότι θα πρόσεχαν κυρίως την εσωτερική τους αγορά αλλά θα συνέχιζαν να εμπορεύονται με, ό με όλες τις χώρες. 3.000 δις δολάρια έχει σήμερα αποθεματικό η Κίνα μετά από τρία χρόνια. Δηλαδή διπλασίασαν τα αποθέματα τους σε δολαρία σε τρία χρόνια. Κύριε Ζαντό, στην τελευταία τοποθέτηση είχατε την απάντηση γιατί δεν θα καταλήξουμε σε καμία σχέση που θα μας βοηθήσει να, μας να προχωρήσουμε τις σχέσεις μας. Στην ίντα πάντα λέγανε είναι η αγορά που αποφασίζει, η αγορά αποφασίζει. Όλοι αυτοί οι οποίοι εμπορεύονται με την Κίνα πήρανε τα κεφάλαια από την Ευρώπη και τα βάλανε στην Κινέζικη αγορά. Και ε, βλέπουμε να υποχωρεί συνέχεια αυτό το ευρωπαϊκό δίκτυο επιχειρήσεων που ε, συγκροτεί ε, τον ευρωπαϊκό χώρο. Τι θα κάνουμε λοιπόν εμείς για να μπορέσουμε να επενδύσουμε ούτως ώστε να διαρθρώσουμε τον βιομηχανικό ιστό στην ευρωπαϊκή επικράτεια και να λύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα για να έχουμε πραγματικές σχέσεις με την Κίνα. Εγώ μέσα στην Ίντα είχα πει ότι ήταν καταχρηστικό να μην λέμε τίποτα όταν μια χώρα η οποία εμπορεύεται και ανατρέπει όλους τους διεθνείς κανόνες εμπορίου για τις εμπριστεχνίες, για την πνευματική διοκτησία. Γιατί, γιατί οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις συμμετέχουν σε αυτή την παροδία. Γιατί παράγουν στην Κίνα και επανεισάγουν προϊόντα τα οποία παράγονται με ευρωπαϊκές εμπρισιτεχνίες και παραβιάζουν όλους τους διεθνούς κανόνες. Η διαφορά μεταξύ κόστους παραγωγής και, κόστους, και, και τιμής πώλησης είναι τεράστια που πραγματικά αξίζει τον κόπο για να πηγαίνουν και αυτό είναι όμως καταστρεπτικό για την απασχόληση, για την βιομηχανία, για, για τις ε, τοπικές κοινότητες. Θα πρέπει λοιπόν εμείς για να μπορέσουμε να διαρθρώσουμε στην επικράτειά μας τις πολιτικές, να έχουμε μία ενιαία φωνή. Ναι πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός, σωστός και ισορροπημένος ανταγωνισμός, όχι ένας ανταγωνισμός που βασίζεται στην απαταιωνία και στην ασέβεια των διεθνών κανόνων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ από τη δική μου πλευρά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή. Έχω. Για την ε, καλή του έκθεση η Κίνα είναι μια πολύ πολύπλοκη ανταγωνίστρια χώρα. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς ε, να έχουμε ελεύθερες ανταλλαγές σε τεχνολογικό και πνευματικό επίπεδο με αυτούς τους όρους. Και σε μεγάλο βαθμό εγώ συμφωνώ με τον προλαλήσαντα συνάδελφο. Δηλαδή θα πρέπει κυρίως να ασχοληθούμε με τη δική μας βιομηχανική πολιτική. Πρέπει τέλος πάντων να αποφασίσουμε να κάνουμε κάτι. Εάν εμείς θέλουμε να αντιμετωπίζουμε την Κίνα ισότιμα με, ως εταίρο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε παγκοσμίως ορισμένα προβλήματα ή θα βλέπουμε απλώς την Κίνα ως μια αγορά για την ανταλλαγή εμπορευμάτων που παράγονται στο εσωτερικό αυτής της αγοράς με, με καθεστώς απόλυτης ασέβειας κοινωνικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πολύ σωστά είπε ο συνάδελφος. Πολλά από τα προϊόντα που αγοράζουμε εμείς εδώ στην Ευρώπη παράγονται στην Κίνα διότι είναι πολύ πιο απλό. Και γιατί η εργασία στοιχίζει πολύ πιο φθηνά στην Κίνα. Δεν υπάρχουν τόσοι κανόνες που πρέπει να γίνονται σεβαστοί. Δείτε όμως και τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές και για αυτές θα πρέπει να επιμείνουμε. Αν εμείς θέλουμε να γίνονται σεβαστοί αυτοί οι κανόνες, δεν μπορούμε να απευθυνόμαστε στους Κινέζους σαν να είναι οι ισότιμοι εταίροι. Πρέπει να τους... Πρέπει να, πουλάμε τα δικαιώ... πρέπει να πουλάμε τις ευρυσιτεχνίες μας, πρέπει να πουλάμε την τεχνολογία, να την αγοράζουν και βάσει συγκεκριμένων όρων να μπορούν να παράγουν. Και χρειαζόμαστε και μια καλή εξωτερική πολιτική. Δεν μπορούμε να το ξεχνάμε αυτό. Δεν θα υπάρξει καμία ανταλλαγή και κανένας ανταγωνισμός ισότιμος εάν δεν έχουμε και τη σωστή εξωτερική πολιτική. Μόνο με αυτόν τον τρόπο εμείς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση και να υπάρχει και μία νομιμότητα για να σταματήσει αυτή η ροή προϊόντων που πουλιούνται με ευρωπαϊκή μάρκα αλλά παράγονται στην Κίνα για να αυξηθεί το κέρδος. Ο κύριος Βίμπερ. Ο κύριος Βέμπερ. Η... Η Αντιπροσωπή Ευρωπαϊκή Ένωση Κίνα, είμαι αντιπρόεδρος της ε, Αντιπροσωπής αυτής, πριν από δέκα μέρες ε, δεχτήκαμε μια αντιπροσωπεία προσώπων ε, του Ευρωπαϊκού Εμπορικού Επιμελητηρίου του Πεκίνου, λέει ο, πρόεδρο, ναι. ο κύριος Βέμπερ. Ε, άνθρωποι οι οποίοι ζουν καθημερινά την οικονομία την κινέζικη. Τι μας λένε οι άνθρωποι αυτοί, μας λένε ότι παρά την τεράστια ευκαιρία την αντιπροσωπεύει η κινέζικη αγορά για τι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει. πρέπει να περιοριστούν από ό,τι παραμένει από την πίτα αυτές οι εταιρείε. Είχαμε την ε, πρόσβαση πριν από 10 χρόνια ε, στον ε, ΠΟΕ, 11 Δεκεμβρίου του 1 συγκεκριμένα προσχώρησε η Κίνα και είχαν γίνει τότε σημαντικές υποσχέσεις, κάποιες από τις οποίες αρκετές πραγματοποιήθηκαν. Είναι η δεύτερη οικονομία σήμερα εκείνα παγκοσμίω, 11% του παγκόσμιου εμπορίου. Και οι επιχειρήσεις της είναι ηγετικές σε πολλούς τομείς, μεταξύ αυτών μελλοντικέ βιομηχανίες όπως ε, φωτοβολταϊκά. Αλλά εξίσου πολλές είναι και οι δεσμεύσεις οι οποίες, τις οποίες η Κίνα αρνείται και δεν εφαρμόζει ποτέ τελικά και αλλάζουν, οι, όπως λέει, οι διάφορες διατάξεις και διοικητικές μεταρρυθμίσεις. Η Κίνα ουσιαστικά παίζει διπλό παιχνίδι, το οποίο είναι πραγματικά παράδεκτο. Τι θα πει αυτό, θα πει ότι ναι, μεν εποφελείται πλήρως του ανοίγματο ε, των δικών μας αγορών, ταυτόχρονα όμως περιορίζει σημαντικά την πρόσβαση των επιχειρήσεών μας στις δικές τους και συγκεκριμένα στους τομείς που θεωρούνται στρατηγικοί για την κυβέρνηση του Πεκίνου. Λίγα παραδείγματα θα σας αναφέρω. 22.000 άδειες ε, τηλεπικοινωνιών από το 2000 και μετά. Από αυτές μόνο οι 14, 14 ε, επί 22.000 πήγαν σε ξένες εταιρείε. Στον τομέα τον τραπεζικό τώρα. Οι μη ε, Κινέζοι ε, τραπεζικοί φορείς κατέχουν λιγότερο του 2% του μεριδίου της αγοράς. Ε, στην οικοδομή, δημόσια έργα, καμία ξένη επιχείρηση δεν έλαβε άδεια για να συμμετέχει ε, στα εργοτάξια την κατασκευή των Ολυμπιακών έργων για την Ολυμπιάδα του Πεκίνου το 2008. Ούτε σε δημόσιες προμήθειες είχαν πρόσβαση οι ξένες Για να μην σα πω γιατί γίνεται και στους σιδηροδρόμους. Πολλά παραδείγματα υπάρχουν και βέβαια όλα αυτά σας κάνουν νομίζω να συνειδητοποιήσετε κάπως τη διάσταση του προβλήματος. Και τελικά φτάνουμε σε εμπορικό έλλειμμα γιγαντίων διαστάσεων που τριπλασιάστηκε και παραπάνω τα τελευταία 10 χρόνια και έχει φτάσει 170 δις ευρώ το 2010. Αυτό είναι το έλλειμμα το οποίο καταγράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις εμπορικές της σχέσεις με την Κίνα. 170 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτό έχει να κάνει και με τη Γερμανία. Και αυτή πλήττεται βλέπουν να μεγαλώνει το χάσμα με την Κίνα το 2010 με εξαίρεση την Ιρλανδία και τη Φινλανδία. Δεν θα μας καταπλήξει λοιπόν το ότι η κοινή γνώμη από αυτές τις συνθήκες ε, φοβάται. Έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντως τη δυνατότητα να παίξει ε, Επίση όρισε το παιχνίδι της Κίνα. Είμαστε εμπορική εταίρη σημαντική. Πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε, να πετήσουμε δυναμικό επαναπροσανατολισμό των ε, συναλλαγών. που σε αυτήν οφείλεται και η κρίση. Θα πρέπει δύο πυλώνες να επικρατήσουν, η ισορροπία και η αμοιβαιότητα. Να υπάρχει fair trade, δηλαδή, εμπορικό, δίκαιο εμπόριο. Και αυτό βασίζεται σε δύο χέσεις, Την αμοιβαιότητα, και την ισορροπία. Δηλαδή ισότιμη ε, συνεργασία. Δεν μπορούμε να ανοίγουμε εμεί τις πόρτες των αγορών μας και να μην κάνουν το ίδιο οι Κινέζοι. Όταν ο Βεν Τζαμπαό ζητάει με φιλικό αλλά επίμονο τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει μια κίνηση, μια χειρονομία καλής θέλησης και να δώσει στην χώρα του το καθεστώς οικονομής της αγοράς πριν την προβλεπόμενη μερομηνία, το 2016 δηλαδή, καιρό είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει μια αποφασιστική στεναρή τάση ό,τι αυτά τα εμπορικά ελλείμματα. Υπάρχουν εργαλεία και μέσα τα οποία έχουμε στη θέση μας και θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε, γιατί αλλιώς πολύ λιγότερο μπορούμε να περιορίσουμε τις ε, τάσεις αναδίπλωσης που βλέπουμε στην κοινή γνώμη στην Ευρώπη. Δεν πρέπει να πέσουμε σε αρνητική αμοιβαιότητα και γι' αυτό θα πρέπει να πιέσουμε τους φίλους και εταίρους μας προς την θετική αμοιβαιότητα, δηλαδή στη βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων των δικών μας στις δικές τους αγορές. Όλοι θα ωφεληθούν, απλά κάποιες φορές πρέπει κανείς ε, να πιεστεί λίγο παραπάνω, να αλλάξει κάποια πράγματα, να μην ε, έχουμε επανάληψη του σεναρίου όπου όλοι θα είναι χαμένοι. Ο κύριος Μπιτικόφερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προτού δημιουργηθεί μια προτεξιονιστική συμμαχία που να περιλαμβάνει όλα τα κομμάτια, όλα τα κόμματα, ε, θα πρέπει να σκεφτούμε αν μια τέτοια στρατηγική θα μπορούσε να είναι επιτυχής και αποτελεσματική. Υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν δικαιολογημένες επικρίσεις, αλλά υπάρχουν και κλισέ. Σε ό,τι αφορά παραδείγματος χάρη την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλοι αυτοί με τους οποίους έχω μιλήσει λένε ότι υπήρξε μια θετική εξέλιξη στην, ε, στην Κίνα και παρόλα αυτά ακούμε μονάχα διαμαρτυρίες και ημωγές για τη θέση της κινέζικης ε, κυβέρνησης που φυσικά έχουν και τη δική τους πλευρά ότι θα πρέπει να υπάρξει και για τις κινέζικες εταιρείες μια προστασία της ιδιοκτησίας τους για να μην ε, τις πάρουν άλλες εξωτερικές εταιρείες. Δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε μια μονάχα μονομερή αντιμετώπιση και να ικανοποιηθούμε με αυτήν θα πρέπει να δούμε την πραγματικότητα. Η λεγόμενη αρχή της αμοιβαιότητος από στατική άποψη είναι ανόητη. Μπορεί κανείς να την έχει και να την κραδένει σαν σύνθημα, αλλά όταν πάει κανείς να δει πώς μπορεί να εφαρμόσει την πράξη αυτή την αρχή, δεν θα πάει πολύ μακριά. Κατά τη δική μου άποψη θα ήταν πολύ χρήσιμο να σκεφτούμε καλύτερα για το θέμα αυτό και να διοργανώσουμε σαν Επιτροπή μια ακρόαση ακριβώ για τα θέματα αυτά που έχουν να κάνουμε με τη σχέση μα και με την Κύριε Ζαντό, θέλετε να επανέλθετε. Με... Βεβαίω. Πρόκειται για μία ενδιαφέρουσα συζήτηση και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στην, βρισκόμαστε στην και όχι στην Ίντα. Είναι πολύ δύσκολο ε, ε, γιατί διαπλέκονται οι κανόνες μεταξύ εμπορίου και βιομηχανίας. Αυτά που είπε η κυρία Χόλ, να διατηρήσουμε ένα μηχανισμό ανταλλαγών, γιατί αυτό είναι υπέρ του καταναλωτή. Ποιο είναι όμως το πρόβλημα είναι ότι ανησυχώντας πια πολύ για τον καταναλωτή ξεχάσαμε τον εργαζόμενο, το κλίμα, τα κοινωνικά δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλαδή όλους εκείνους, όλες εκείνες τις θεμελίες που βασίζουν μια διεθνή κοινωνία. Πρόκειται για την κρίση μιας ίδιας λογικής, δηλαδή που για να εξυπηρετήσει, ισχυριζόμενη ότι εξυπηρετεί τον καταναλωτή, οδηγήσαμε τους σε τέτοιες καταστάσεις ανταγωνισμού που δεν ξέρουμε πια τι κάνουν οι οικονομίες μας και οι κοινωνίες μας. Για την αμοιβαιότητα. Εγώ καταλαβαίνω την ιδέα ότι οι Κινέζοι εκμεταλλεύονται μια πολύ διευκολυμένη είσοδο στις αγορές μας και των ε, ε, δημοσίων αγορών και των διαγωνισμών και δημοπρασιών. Εμείς θα μπορούσαμε να αποκαταστήσουμε την κατάσταση λέγοντας ότι οι Κινέζοι θα έπρεπε να μας προσφέρουν αντίστοιχα αυτό το οποίο εμείς τους προσφέρουμε στις αγορές μας. Τι θα γινότανε. Αν εγώ δω τι γίνεται πολυμερός σήμερα. Η ΔΟΕ λειτουργεί άσχημα οι διαπραγματεύσεις ε, για το κλίμα είναι στάσιμες, ε, ε, βλέπουμε ποια είναι η λογική των Κινέζων και των ΙΠΑ για το κλίμα, ανθρώπινα δικαιώματα, θεωρώ ότι το κινέζικο καθεστώς είναι ένα καθεστώς το οποίο δεν εξελίσσεται γρήγορα για την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων και χρησιμοποιεί τα κοινωνικά δικαιώματα υπέρ του ανταγωνισμού ε, των ε, ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Δείτε το νόμισμα που δεν είναι θέμα της Ήτρε. Αλλά το G20 είναι εντελώ αναποτελεσματικό να, να, διαχειριστεί την όλη ιστορία του κινέζικου νομίσματος. Λοιπόν, κοιτάστε, αν το G20 ή G8 είχαν αποφασίσει ε, κάτι το ουσιαστικό ε, θα γινότανε. Όχι γιατί ο Σαρκοζή πάει και, και προεδρεύει τις ε, διασκέψεις κορυφής και είναι μόνο λόγια χωρίς έργα τελικά. Αυτή τη στιγμή παραμένει μία μεγάλη παγκόσμια αγορά ε, θα πρέπει να παραμείνει και χωρίς εδώ να θέλω εγώ να, ε, να, να, να, να παίξω τον, ε, πάνω στην ευρωπαϊκή Ενωτερότητα, αλλά πρέπει να επιβάλλουμε τους όρους σεβασμούς Θα πρέπει η Ευρώπη να θέσει ισχυρούς κανόνες και για το νόμισμα κοινωνικά δικαιώματα περιβάλλον. Ο κύριο Σενέ, νομίζω και κάποιος άλλος θέλει να θέσει ένα σύντομο ερώτημα, αλλά πάρα πολύ σύντομο. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο, κύριε Πρόεδρε. Υποσχέθηκα να είμαι πολύ σύντομο. Εμείς εδώ είμαστε ένα κοινοβούλιο με διαφορετικές γνώμες που εκφράζονται. Και αυτό είναι και η δύναμή μας, η διαφορά. Και ξέρουμε να συζητάμε. ακόμη και αν έχουμε διαφορετικές απόψεις. Λοιπόν, ο κύριος Μπουτιχόφερ θέλει να προχωρήσει σε μία ακρόαση εμπειρογνωμόνων. Τον παρακαλώ λοιπόν όμως να είναι με τα πόδια... Να είναι με τα πόδια στη γη. Ο κύριος Βέμπερ. Για τον κύριο... Η αμοιβαιότητα δεν είναι βλακεία. Τι είναι η αμοιβαιότητα. Αν οι Κινέζοι έχουν δικαίωμα να κατασκευάσουν ένα τμήμα του αυτοκινητοδρόμου μεταξύ Βαρσοβίας και Βρόκλαβ, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα, έχουν, θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να κάνουν την ίδια δουλειά στην Κίνα. Αν οι Κινέζοι θέλουν να αγοράσουν τη Volvo ή τη Saab, τότε και οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να κοιτάξουν να κάνουν τέτοιο πράγμα στην Κίνα στις αυτοκινητοβιομηχανίες. Σήμερα είναι αδύνατο στην Κίνα ένας αυτοβιο... μια αυτοκινητοβιομηχανός δεν μπορεί να κατέχει πάνω από το 50% το οποίο θέλουν να το μειώσουν σε 49% τώρα στην Κίνα. Να δείξουμε λοιπόν κι εμείς όμως ότι μπορούμε να κάνουμε αυτό που κάνουν οι Κινέζοι και οι Αμερικάνοι, δηλαδή να φούμε. Να δείξουμε ότι ξέρουμε να φούμε. Λοιπόν, πρόκειται για μια καταπληκτική αγορά, δεν θέλω να τους γυρίσουμε την πλάτη, αλλά αυτό χωρίς απλοϊκότητα και με μια κάποια δυναμική και ρεαλισμό. Μερσή λέει ο πρόεδρος, 13 Οκτωβρίου την 5η είναι στη μία η ώρα είναι η προθεσμη για τις τροπολογίες. Ερχόμαστε στο επόμενο θέμα που είναι η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας. Ο κύριος έχει το λόγο. Σε ό,τι αφορά την περιφερειακή διάσταση της πολιτικής γειτονίας, θεωρώ ότι αυτή είναι μία από τις προτεραιότητες αυτής της πολιτικής τα επερχόμενα χρόνια. Θέλουμε να ενισχύσουμε και τις δύο διαστάσεις και την ανατολική και την νότια πολιτική γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να εξασφαλίσουμε μια ισορροπία μεταξύ των δύο αυτών πτυχών της πολιτικής. Είναι δύο πτυχές της ίδιας πολιτικής για μας. Η τομεακή συνεργασία με τις χώρες αυτές είναι πάρα πολύ σημαντική και όχι μονάχα η ενεργειακή πολιτική. Μας ενδιαφέρει να αναπτύξουμε νέους ενεργειακούς φορείς και επίσης να συνδέσουμε την ενεργειακή πολιτική με την πολιτική αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Η συνεργασία για τη Μεσόγειο και για τα θέματα τροφοδοσίας με το φυσικό αέριο. Όλα αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικά θέματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι στοιχεία που μπορούν να ενισχύσουν την σταθερότητα και φυσικά και την ασφάλεια εφοδιασμού σε ενέργεια. Ποια είναι λοιπόν τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε για να χρησιμοποιήσουμε για να ενσωματώσουμε την ενεργειακή πολιτική με την πολιτική εμπορίου και την πολιτική γειτονία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σαφές ότι θα πρέπει να εμπλακεί σε μια σαφέστερη, σε μια στενότερη συνεργασία στον τομέα τη ε, καινοτομίας και της έρευνας να δημιουργηθεί ένας κοινό χώρος έρευνας και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της διαβίου εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η Κομισιόν θέλει να υπάρξουν συγκεκριμένα κονδύλια τα οποία θα προσδιοριστούν 1022 ευρώ συγκεκριμένα, εκατομμύρια μάλλον ευρώ. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν και μια υποστήριξη που θα υποστηρίξει αυτούς οι οποίοι παίζουν ηγετικό ρόλο στις αλλαγές στις χώρες του Νότου και της Ανατολής. Πρέπει επίσης να υπάρξει η αιρεσιμότητα και να διαφοροποιηθεί και η προσφορά μας και σε οικονομικούς αλλά και σε κοινωνικούς όρους θα πρέπει όλα να βασίζονται στην πραγματική θέληση προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπό πολωνική Προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κομισιόν θα πρέπει να ξεκινήσει τις προετοιμασίες για να μπορέσουμε να έχουμε ενισχυμένη συνεργασία για τα δυνητικά επερχόμενα κράτη-μέλη. Χρειάζεται λοιπόν μια καλύτερη συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής γειτονίας, η οποία θα πρέπει να εστιάσει και περισσότερο στα ωφέλη τα οποία μπορούν να προκύψουν για τους γείτονές μας προς Νότον και προς Ανατολή, εάν συμμορφωθούν με τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Η Αραβική Άνοιξη έδειξε ότι η Ευρώπη πρέπει να αναθεώρησε την εξωτερική της πολιτική και να στηρίξει τις πραγματικές δημοκρατίες. Στηρίζουμε τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, αλλά αυτό θα πετύχει μόνο αν αναπτύξουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική η οποία πραγματικά θα υποστηρίζει ένα αλληλέγγυο οικονομικό μοντέλο που θα μπορεί να περιορίσει τις σημαντικές κοινωνικές ανισότητες και να δημιουργήσει απασχόληση. Γι' αυτό και η γνωμοδότηση της ΣΥΤΡΑ για το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντική κατά την άποψή μου. Διάβασα προσεκτικά το πολύ καλό σχέδιο γνωμοδότηση του εισηγητού και φυσικά συμφωνώ μαζί του ως προς το ότι ο τομέας που σίγουρα έχει τη μεγαλύτερη δυνατότητε όθηση ό,τι αφορά την οικονομική ανάπτυξη, για τι γειτονικέ χώρε μιλάω, είναι ο τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Βέβαια, για να γίνει πράξη αυτό, θα πρέπει να στηρίξουμε τα έργα εκείνα τα οποία ε, παρέχουν νέες πηγές ε, πόρων ε, απασχόλησης, ενισχύουν τις υποδομές δικτύων των γειτόνων μας και επιτρέπουν στις χώρες αυτές να αναπτυχθεί ένας νέος βιομηχανικός τομέας και συμφωνώ και από αυτού του σημείου με τον εισηγητή στον τομέα τώρα της έρευνας. Κάνει σύντομη αναφορά σε αυτό το θέμα ο εισηγητής. Η ομάδα μας είναι πεπισμένη ότι η όθηση για αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία εργασιακών ευκαιριών θα συμβαδίζει και με τον, τη δημιουργία ενός ε, ενιαίου χώρου γνώσεων. Ξέρετε ότι η Συμφωνία Σύνδεσης αυτή είναι η καλύτερη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε ε, και θα πρέπει να υπάρχει η διαδικασία αυτή στις χώρες οι οποίες βρίσκονται σε φάση μετάβασης στον τομέα των γνώσεων της έρευνας, ό,τι αφορά τη συνεργασία των επιχειρηματιών και αυτό είναι σημαντικό για να σημειώσουμε πρόοδο στον τομέα των ελεύθερων συναλλαγών θα πρέπει να έχουμε μια κανονιστική σύγκληση και να παρέχουμε και χρήσιμες πληροφορίες για τις ε, εμπορικές σχέσεις και τις επενδυτικές ευκαιρίες των επιχειρήσεων, ιδίω των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτή είναι η λόγη που θα κάνουν την ομάδα μου να επικυρώσουν πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες όπως ο Ευρωμεσογειακός Μηχανισμός Διευκόλυνσης του Εμπορίου ή εμβληματική πρωτοβουλία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο πλαίσιο της οριζόντιας σύνθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. <clears throat> Η Κομισιόν θα ήθελε να παρέμβει. Κύριε Μανκεβίτς, θέλετε να πείτε κάτι ακόμα. Όχι. Εντάξει, είμαστε στην ώρα μας λοιπόν. Μπορούμε να κλείσουμε και αυτό το σημείο της ημέρας της διάταξης τουλάχιστον προς το παρόν. 27 Σεπτεμβρίου στις 12 η ώρα είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες. Έχουμε κλείσει και αυτό το σημείο, το σημείο 15. Έχουμε ένα-δύο λεπτά για τις ε, ψηφοφορίες. Ένα-δύο λεπτά. Στις 10 ακριβώς ξεκινάμε. Okay. Perhaps we can start again. Oh. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Όλοι στο πλοίο. Έχετε τις κάρτες ψηφοφορίας σας. Το μηχάνημα δουλεύει. Εντάξει, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Η πρώτη ψηφοφορία λογικά Συμμετοχή επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων στι έμεσε δράσει βάσει του προγράμματο πλαισίου τη Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομική Ενέργεια. Τέσσερι εκθέσει του κυρίου Μπριζίνα, αλλά είναι χωριστέ. Παρακαλώ, να προσέξετε τη σωστή σειρά για να μην τα, κάνουμε, να μην τα μπερδέψουμε. Μάλιστα. Όλοι έχετε κάρτες. Τις κάρτες ψηφοφορίας. Όλοι έχουν τις κάρτες Κάποιος έχει πρόβλημα. Έκθεση Μπρεζίνα η πρώτη. Άρθρο 4. Ψήφι υπέρ. Κατά. Χες. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 2. <clears throat> Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 14 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Έχετε πρόβλημα Giles. Ποια είναι η έκθεση από τις τέσσερις εκθέσεις Βρεσίνα που ψηφίσουμε. Αν μπορείτε να με βοηθήσετε κιόλας. Δεν αντιστοιχεί στη σειρά που έχω εδώ μπροστά μου. Η πρώτη έκθεση είναι αυτή που φέρει τον αριθμό 73. Συμμετοχή πανεπιστημίων ερευνητικών κέντρων στο πρόγραμμα πλαίσιο της ε, ε, Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας. Εντάξει, το καταλάβατε. Δεν θα ξαναρχίσουμε από την αρχή βέβαια. Εντάξει. Τροπολογία 14. Πρώτο τμήμα κατά αποχές εντάξει δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή 16, 17, 18, 20 και 21 unblock ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 5. Υπέρ. Έχετε πρόβλημα, κυρία Φόρτ. Ποιο είναι το πρόβλημά σας. Ο κατάλογος ψηφοφορίας μας δεν φαίνεται να αντιστοιχεί με αυτά τα οποία ψηφίζουμε. Καθόλου. Είναι το 73 που ψηφίζουμε. Όχι, λέει ο πρόεδρος. Κύριε Μπρεζίνα, μήπως μπορείτε να μας βοηθήσετε εσείς. Sind wir soweit? Εντάξει. μία-μία τις ε, ψηφοφορίες με τη σειρά που τις έχουμε στην μέση διάταξη. Ακολουθούμε τη σειρά που υπάρχει στην μέση διάταξη. Έχει πολύ ωραία νουμεράκια. Δεν ξέρω αν έχετε δυσκολία να τα, διαβάσετε. Είναι για να σας βοηθήσουν. Μην προσθέσετε όμως τους αριθμούς γιατί θα, θα μπερδευτείτε. Εντάξει. Ωραία. Είμαστε τώρα στις αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 8. Υπέρ κατά αποχές δεκτή 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά πάντα άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας Εγκρίνεται. Ο Κλοντ Τούρμες θέλει. Και εσύ έχεις τον μπερδεμένο το λάθος κατά. Εγώ θα ψήφισα κατά γιατί δεν έχω την κάρτα μου, ε, οπότε πρέπει να προσθέσουμε μία ψήφο τους κατά. Και εσείς, υπέρ ή όχι. Και εγώ δεν είχα κάρτα, αλλά είμαι υπέρ, λέει η κυρία Μαδουρέλ. Ωραία. Δύο ακόμα παραπάνω υπέρ και μία ψήφος παραπάνω κατά. Επόμενη ψηφοφορία Μπρεζίνα. Όπως στην, τροπολο... στην μέση διάταξη. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ. Η 16 είναι το 16, λέει ο πρόεδρος στα αγγλικά. Είναι η τροπολογία 16 είναι το έγγραφο που τελειώνει σε 0073, αν έχετε κάποιο πρόβλημα. Μα δεν γίνεται στη σωστή σειρά που έχουμε στον κατάλογο ψηφοφορίας. Είναι, μας κάνει πολύ μεγάλη δυσκολία να παρακολουθήσουμε τι γίνεται. Έχουν το δικό τους κατά. Αν η ομάδα σας έχετε κάνει διαφορετικούς καταλόγους ψηφοφορίας, εγώ δεν φταίω. Εγώ ακολουθώ τη σειρά των καταλόγων ψηφοφορίας που βρίσκεται στην ημέρησια διάταξη. Μόνο έτσι μπορεί να λειτουργήσει κανείς για να μην έχουμε απόλυτο χάος. No, no, no, please. Now uh, first. your, uh, because it is uh, voting list of committee, official voting list of ITRE and your... Είναι η επίσημη λίστα της Επιτροπής ITRE αυτή που έχουμε. Τι να σας πω, όποιος δεν είναι σίγουρος σας κάνει ό,τι κάνω εγώ. Δεν φταίτε εσείς κύριε Μπρεζίνα, ακολουθούμε ακριβώς την ημερήσια διάταξη και την ε, λίστα που έχει προετοιμάσει η γραμματεία της Επιτροπής. Ο Τζάιλ Σέτσιτσεσταν και πάλι και ο κύριος Τόιρερ μετά. Εγώ ευχαρίστως να ακολουθήσω ό,τι κάνει ο κύριος Μπρεζίνα. Αλλά νομίζω ότι το πρόβλημα είναι η γραμματεία που παρέλειψε να μας στείλει την επίσημη λίστα ψηφοφορίας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εξού και η σύγχυση. Φαίνεται ότι και άλλες πολιτικές ομάδες αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, άρα μυρίζομαι ότι φταίει η γραμματεία. Λοιπόν, ας πούμε ότι φταίει η γραμματεία, ζητώ συγγνώμη τη γραμματεία, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να προχωρήσουμε. Εντάξει. Εγώ δεν έχω δει τον κατάλογο. Εγώ έχω την τελική ευθύνη και προχωράμε. Είναι το έγγραφο 0073. Σύμφωνοι. Το έγγραφο που τελειώνει σε 0073 στο τέλος. Πρώτη ψηφοφορία έχει γίνει. 16. Τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές εντάξει. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 17 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ, κατά αποχές υπέρ πάλι, γιατί 19 υπέρ, υπέρ, υπέρ, υπέρ, κατά Αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Χωριστή ψηφοφορία για την 20. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Χες. Απορρίπτεται. 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 1 υπέρ <clears throat> κατά αποχές εγκρίνεται 4 όχι όχι συγγνώμη εκπίπτει 23 έχει αποσυρθεί 24 υπέρ 24 24 23 έχει αποσυρθεί. 24. Υπέρ. 24. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχέ και αυτή εγκρίνεται. 26. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά άρχεται. Close. No. Closed. Πέρας. And adopted. Εγκρίνεται. Τρίτη έκθεση Μπριζίνα. 0074. Όλο και καλύτερα τα πάμε. 3 υπέρ. Κατά. Αποχέ απορρίπτεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 12 αποσύρθηκε. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 14 <clears throat> <clears throat> με προφορική τροποποίηση υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Διαδικαστική παρέμβαση. Είναι το decommissioning. Δεν το έχω αποσύρει. Εμένα λέει ο κατάλογος μου ότι την έχετε αποσύρει, σας ευχαριστώ όμως. Προφανώς θα πρέπει να ψηφίσουμε. 12 ψηφίζουμε υπέρ. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίθηκε. 15. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. 16. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 17 εκπίπτει. 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Εκπίπτει 19, 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ένα του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο τμήμα υπέρ πρώτο τμήμα της 24 ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Το έλκα έχει ένα που περισσεύει. Μία κάρτα πρέπει να βγει. Εντάξει. Και το αποτέλεσμα είναι α, εγκρίνεται λέει ο πρόεδρος. Συγγνώμη, απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δύο του εισηγητή υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 25 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 26. Στο δεύτερο τμήμα υπήρχε μια προφορική τροποποίηση, λέει ο κύριος Τούρμες. Εγώ είμαι κατά αυτής της προφορικής τροποποίησης. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να πούμε και το δεύτερο τμήμα με την προφορική τροποποίηση ότι πρέπει να ψηφίσουμε. Α, τώρα κατάλαβα, δεν θέλετε. Οι πράσινοι δεν δέχονται την προφορική τροποποίηση. Επομένως η τροπολογία δεν είναι παραδεκτή. Δεύτερο τμήμα χωρίς την προφορική τροποποίηση. Συμφωνεί. Εντάξει. χωρί την προφορική τροποποίηση που δεν τη δέχονται οι πράσινοι. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 26 <clears throat> υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 6 υπέρ κατά αποχές δεκτεί 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρας. Ένας από το ΕΛΚ περισσεύει. Βγάλτε μια κάρτα. Εντάξει. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. Τέταρτος Μπρεζίνας. 0.72. Ξεκινάμε με την τροπολογία 9. Κυρία Χολ, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Θέλω παρακαλώ να σημειώσετε ότι έχω μια προφορική τροπολογία. Συγκεκριμένα, νομίζω, επί της τροπολογίας 23. Θα το βρω, θα το βρω και θα επανέλθω. Πέστε μου όταν φτάσουμε εκεί, λέει ο πρόεδρος. 9. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ένα. Υπέρ, κατά, αποχές δεκτή 31 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή 32 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 3 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή 33 και 34 μαζί ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται, συγγνώμη, 35 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ. Η 6 είναι ταυτόσιμη με τη 36. 37 είπα, λέει ο πρόεδρος. 37 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 30... 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Σαράντα δύο τώρα. Σαράντα δύο. Και οι οκτώ. Συγγνώμη. 8 προϋπολογισμών υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα 42 όμως. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 43. Κυρία Χόλ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να προτείνω μια προφορική τροπολογία. Ουσιαστικά πρόκειται για μια αλλαγή γλωσσικού ήχους έχει να κάνει με, το, με τη μετάφραση στο Tabling Office. Τροπολογία και της κυρίας Βαλιάν θα πρέπει να λέει ότι οι πυρηνικέ δραστηριότητες στο πλαίσιο του ΚΚ ερευνών που έχει να κάνει με το nuclear safety στα αγγλικά και όχι security. Nuclear safety, όχι nuclear security. Στα ελληνικά είναι η ίδια λέξη. Δεν βλέπω καμία αντίρρηση. Μπορούμε να ψηφίσουμε λοιπόν με αυτή την τροποποίηση 43, με αυτή την προφορική δια, διευκρίνηση υπέρ, κατά, απόχες εγκρίνεται. 44 υπέρ, κατά, απόχες εγκρίνεται. 45 ψήφι υπέρ, κατά, απόχες εγκρίνεται. 46 υπέρ, κατά, απόχες εγκρίνεται. 47 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53 και 54 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 56 και 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 59 υπέρ κατά αποχές δεκτή 60 σαν προστίκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 63 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 66 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 67 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 εκπίπτει, 17 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 23 24 λέει ο πρόεδρος 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2 του προϋπολογισμού υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ, κατά αποχές συγκρίνεται τελική ψηφοφορία άσχετη η ψηφοφορία τρικά. πάλι ένας από το ΕΛΚ περισσεύει εγκρίνεται εντάξει ευχαριστώ σημείο 20 τώρα ε, συγχαρητήρια κύριε Μπρεζίνα 4-0 με ένα σπάρο 4 τριγώνια ε, οδηγός χάρτης για ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο, τροπολογία 1, συμβαστική, κατά, δεκτή, συμβαστική 2, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 8, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 3, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 15, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 16, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 με τροφορική τροποποίηση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σα... Τι θέλετε, τι να ελέγξουμε. Την 38, μάλιστα. Με προφορική τροποποίηση καθυστερήσατε, αλλά καλή αργά παραποτέ. Πάμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ε, ναι, κρίθη. Με μια μικρούλα πλειοψηφία. 39 την ψηφίσαμε, 41 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 μετροφορική τροφορική τροποποίηση. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται κύριε Κάλς. Υπήρξε μια υποστήριξη από όλους, ομοφωνία. Τελευταίο σημείο. Ανοιχτό διαδίκτυο και διαδικτυακή ουδετερότητα στην Ευρώπη πρόκειται για μία προφορική ερώτηση μονάχα. Αυτό είναι το εύκολο κομμάτι. Ποιο ψηφίζει αυτή την προφορική ερώτηση. Υπέρ. Κανείς. Α, ωραία. Κατά. Ερώτηση με έτοιμο προφορικής απάντησης στο όνομά μου. Υπέρ κατά Δεν έχουμε τροπολογίες εδώ. Είναι πολύ δύσκολο ερώτημα το αν θα θέσουμε προφορική ερώτηση όχι. Άμα σας ξεπερνάει εντάξει θα το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Παρ' όλα αυτά ποιος θέλει να υπερψηφίσει. Κατά. Αποχές. Ε, ομόφωνα είναι κρίθη. Ωραία. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ τα μάλα. Το επόμενο σημείο σας ευχαριστώ για τις ψηφοφορίες και ερχόμαστε τώρα στο θέμα χάρτη πορεία για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επίπεδων ανθρακούχων εκπομπών μέχρι το 2050 θέλει ο Θεός. Ο εισηγητής είναι ο κύριος Πυριλό. Είναι ο πρώτος που θα λάβει το λόγο. Όσοι θέλουν να φύγουν παρακαλώ να φύγουν ηρέμος, ησύχος. Αν θέλετε να μείνετε εδώ πέρα, αυτό είναι ακόμα πιο συγκινητικό. Να βοηθήσετε τον κύριο συνάδελφο, άμα θέλετε όμως να κάνετε πηγαδάκια, έξω σας παρακαλώ. Κύριε Πυρίλα, λό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η ανακοίνωση της Επιτροπής ε, για τον Οδικό Χάρτη 2050 είναι μία από τις ε, πιο σημαντικές εργασίες μας ε, των επομένων μηνών και που θα οδηγήσει ακριβώς σε πολιτική συζήτηση. Εμείς πρέπει να φανταστούμε σενάρια για τη μείωση των εκπομπών τα επόμενα 40 χρόνια. Στο σενάριο το οποίο έχει φανταστεί η Κομισιόν ζητείται σημαντική προσπάθεια στον τομέα παραγωγής ηλεκτρισμού που πρέπει να μειώσει κατά 50% τις εκπομπές της. Ζητείτε, για την ακρίβεια ζητείται να μειωθούν οι εκπομπές ε, κατά 80%. Πρέπει να φανταστούμε λοιπόν συνολικά όλο το κοινωνικο-οικονομικό σύστημα, όχι μόνο το σύστημα παραγωγής ενέργειας. Πρέπει να φανταστούμε καλύτερη χρήση της επικράτειας και της διαχείρισης των πόρων, των ενεργειακών πόρων. Οι επιλογές τις οποίες καλούμεθα να κάνουμε πρέπει να είναι ακόμη πιο διαρθρωμένες και αυτό λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι ιδιώτες και οι επενδύσεις λόγω της οικονομικής κρίσης. Αληθεύει ότι μετά από μια κρίση μπορούμε να έχουμε αναπτυξιακές ευκαιρίες, αλλά τι, αν ο στόχος 2050 έχει να, ε, παραμένει να μειώσουμε κατά 80 έως 95% τις εκπομπές φυσικού αερίου, ε, τις εκπομπές αερίων που οδηγούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου πρέπει να βρούμε δράσεις και πολιτικές δίνοντας ρεαλιστικές και σοβαρές κατευθύνσεις κυρίως εφικτές που θα μπορέσουν να βοηθήσουν και στην ενεργειακή ασφάλεια της ευρωπαϊκής οικονομίας. Έχουμε πολλές δυνατότητες και πρέπει να τις αναλάβουμε ταυτόχρονα, διότι καμία από μόνη της δεν επαρκεί για να μειωθούν επαρκώς οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος. Έτσι όπως λέω στη γνωμοδότησή μου έχουμε προτεραιότητες επί των οποίων πρέπει να παρέμβουμε. Έναν κεντρικό ρόλο θα πρέπει να τον έχει η έρευνα για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τεχνολογίες με χαμηλές εκπομπές, αποθήκευση της ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αύξηση της αποδοτικότητάς του είναι σαφές ότι θα πρέπει στο νέο ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα από ό,τι σε άλλους τομείς στον τομέα της ενέργειας. Η έρευνα στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο επίσης πρέπει να ενισχυθεί. Όλοι γνωρίζουμε ότι το 20% ε, ενεργειακής αποτελεσματικότητας που ορίζει η Ατζέντα 2020 δύσκολα θα προσεγγιστεί. Πρέπει λοιπόν να συγκεντρώσουμε όλες μας τις προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα πρέπει να έχουμε target ιδιαίτερα δεσμευτικά. Πρέπει να επιμείνουμε στην ενεργειακή αποτελεσματικότητα των κτηρίων, με φοροαλαπαλλαγές, επενδύσεις και παρεμβάσεις. Ε, θα πρέπει να επέμβουμε επίσης υπέρ των εφιών μετρητών ε, και στα συστήματα διανομής. Μεταξύ της ενεργειακής βεντάλιας που θα πρέπει να εξετάσουμε θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τους διάφορους τομείς. Από το 2013 θα αρχίσουν να επιβαρύνονται ορισμένοι τομείς. Οι άμεσες εκπομπές και η περικοπή αυτών των εκπομπών στις, ε, ε, από, ε, στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ή η φορολόγηση τους οδηγούν σε μία στρέβλωση του ανταγωνισμού. Πρέπει να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε τους πολιτικούς στόχους της roadmap ενισχύοντας και το σύστημα των επενδύσεων και των νέων τεχνολογιών για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα και αυτάρκεια. Χρειάζεται να έχουμε μία ρυθμιστική σαφήνια για τους στόχους που θέλουμε να προσεγγίσουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βιδάλ ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Γνωρίζουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση μικρόφωνο είναι. Έχει προβεί σε μια μονομερή απόλυτη δέσμευση για τη μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα κατά 20% μέχρι το 2020 σε σχέση με τα επίπεδα του 90, του 1990. Το Συμβούλιο αποφάσισε να συμπληρώσει τους στόχους αυτούς με ένα πολύ πιο φιλόδοξο μεσοπρόθεσμο στόχο για το 2050 Ο στόχος αυτός είναι μεταξύ του 80% και του 95% μέχρι το 2050. Άρα υπάρχει μια ξεκάθαρη ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να συντονίσει όλες τις δράσεις της, όλες τις πολιτικές της προς αυτό το μεσοπρόθεσμο στόχο. Και βέβαια ο δικός αυτός χάρτης είναι ένα πολύ καλό βήμα προς τα εμπρός για την επίτευξη του στόχου αυτού. Παρ' όλα αυτά όμως αυτά πρέπει ο δικός ε, χάρτης να εκπροσωπεί μια σωστή οικονομική πολιτική ε, κρίση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όλο αυτό θα επηρεάσει τους στόχους αυτούς. Υπάρχουν δύο ουσιαστικά σημεία που θα πρέπει να έχουμε κατά νου. Το πρώτο είναι ότι βρισκόμαστε εν μέσω μιας πάρα πολύ σκληρής οικονομικής κρίσης που πόρα απέχει του να ε, πλησιάζει προς το τέλος της. Και το δεύτερο σημείο είναι ότι είμαστε απομονωμένοι, είμαστε μόνοι μας. Δεν εφαρμόζει κανένας άλλος ε, μέτρα περιβαλλοντικά, μέτρα αηφορίας. Κάποιες χώρες πράγματι προσπαθούν κάπως ε, να ανακτήσουν λίγο χαμένο έδαφος, κάποιες αναδεόμενες οικονομίες όπως η Βραζιλία, η Κίνα, με καλά αποτελέσματα. Δεν θα πρέπει όμως να το ξεχνάμε ότι προς το παρόν είμαστε αρκετά απομονωμένοι. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να κάνω λίγες παρατηρήσεις. Πρώτη παρατήρηση. Πρέπει να βασιστούμε στις επιχειρήσεις μας, στον ιδιωτικό μας τομέα, ώστε να έχουμε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα σε αποδεκτά επίπεδα. Να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και για να γίνει αυτό πρώτον πρέπει να προσελκύσουμε κεφάλαιο. Αυτό αποτελεί ειδικότερα την ευθύνη των πολιτικών που θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα καλό πολιτικό και ρυθμιστικό πλαίσιο και κατά δεύτερον θα πρέπει να επιτρέψουμε στην ελεύθερη οικονομία της αγοράς να μπορεί πράγματι να λειτουργεί ελεύθερα και να είναι μακροπρόθεσμα και προβλέψιμη. Σε ό,τι αφορά την ενέργεια τώρα που είναι και ο βασικός παράγοντας που θα μας οδηγήσει σε μια οικονομία με χαμηλές κομπές ε, διοξυδίου του άνθρακα. Η ενεργειακή αγορά λοιπόν έχει να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο και πρέπει να υπάρχει και ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού για να μπορέσει η αγορά αυτή να εκπληρώνει τους ε, προσδοκόμενους στόχους ε, και στο σύστημα ETS για την ανταλλαγή δικαιωμάτων ε, εκπομπών. Οι αρχικοί κρατών και κυβερνήσεων φέτος επανέλαβαν για μια ακόμη φορά το ότι το ETS θα πρέπει να είναι το βασικό εργαλείο για μια οικονομία χαμηλών επίπεδων εκπομπών άνθρακα όμως η απανθρακοποίηση, αν θέλετε αυτή τη στιγμή, βασίζεται κατά κύριο λόγο στι επιδοτήσει, οι οποίες όμως στρεβλώνουν την αγορά. Ποιο είναι το πρόβλημα. Αν ε, το δούμε υπό όρους μακροπρόθεσμης στρατηγικής. Οι επιχειρήσεις, οι επιλογές που θα κάνουν δεν μπορούν να βασίζονται μόνο στι επιδοτήσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αυτό στρεβλώνει πλήρω την αγορά. Είναι δε άκρος αρνητικό για ένα μακροπρόθεσμο όραμα. Αληθεύει ότι το ETS ίσως πρέπει να βελτιωθεί, ιδίως ό,τι αφορά τη διαφάνεια. Είναι πάντως πολύ σημαντικό οι επιδοτήσεις που στρεβλώνουν τις τιμές του άνθρακα να αρθούν. Αν άρουμε βέβαια τις επιδοτήσεις, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε τραυματικά βραχυπρόθεσμα ε, αποτελέσματα και επιπτώσεις. Αλλά Τούτου λεχθέντος πρέπει να έρθουν μακροπρόθεσμα επιδοτήσεις. Το να περάσουμε λοιπόν από ένα σύστημα επιδοτήσεων σε ένα άλλο σύστημα είναι κάτι δύσκολο ως εγχείρημα. Πρέπει να το σχεδιάσουμε προσεκτικά και δεν θα πρέπει να μας απασχολούν ε, κοντόθωρες ε, κομματικές ε, σκέψεις. Σίγουρα θα πρέπει να σκεφτούμε και τις απαραίτητες στρατηγικές αποφάσεις. Και θα πρέπει να επενδύσουμε σε έρευνα για την ε, μείωση των εκπομπών άνθρακα και θα πρέπει να προσαρμόσουμε και το εργατικό δυναμικό στις νέες δεξιότητες και στις νέες ανάγκες. Πιστεύω λοιπόν στην ανάγκη νέων μακροπρόθεσμων προγραμμάτων όπως είναι το CCS ε, ή ε, το ITER. E για την ε, συγκράτηση αποθήκευση άθρακα και το ίτερ για τη θερμοπυρηνική σύνδεξη. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και αργότερα και για την ενεργειακή απόδοση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την διαλειτουργικότητα και την ε, διασύνδεση του δικτύου. Εάν δεν αρχίσει να υπάρχει διασύνδεση των δικτύων, αν δεν μπορούμε να τα προσαρμόσουμε τα δίκτυα στις αγορές, ε, στο ενεργειακό μείγμα, τότε το μέλλον της ενεργειακής ασφάλειας φαίνεται λίγο ζωφερό. Και σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, ιδίως ε, σε δεινούς καιρού, σαν τους σημερινούς, είναι ένα πολύ λεπτό αλλά πάρα πολύ κρίσιμο θέμα. Η πράσινη ενέργεια είναι δαπανηρή ενέργεια και όπως είπα είμαστε απομονωμένοι προς το παρόν. Άρα θα πρέπει να γίνει μια ρεαλιστική αντιμετώπιση των εξόδων από τις αγορές και υπολογισμός τους και να προωθήσουμε ταυτόχρονα και τη θέση, ε, τις θέσεις εργασίας στην πράσινη οικονομία, την έρευνα και την ανάπτυξη. Είμαι της άποψης, όπως και πολλοί από εσά, ότι η έκθεση αυτή είναι επίκαιρη και έχει έρθει η στιγμή να βρούμε πρακτικές αποδοτικές λύσεις για να, ε, για να πετύχουμε τους στόχους μας στην οικονομία στις παρούσες δύσκολες συνθήκες. Από ό,τι άκουσα από τον κύριο Πυρίλο, πραγματικά έχω σχηματίσει την καλύτερη εντύπωση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φράνκο, αλλά θέλω να κάνω μια μικρή παρατήρηση. Σας παρακαλώ να προσπαθήσουμε να είμαστε λίγο σύντομοι γιατί έχουμε αρκετές εκθέσεις σήμερα. Κύριε Φράνκο, έχετε το λόγο. Χωρίς μικρόφωνο. Oh, ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Θεωρώ ότι η Κομισιόν το παρατράβηξε με τις λεπτομέρειες. Η φιλοδοξία δεν την αμφισβητεί κανένας, αλλά ε, εδώ τα, η λεπτομέρεια είναι τέτοια που περισσότερο μοιάζει με, με, κανονισμό παρά με οδηγία, με, δίνει κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να κρατήσουμε τη γραμμή που είχαμε ορίσει ε, την άνοιξη του 2011 στο Συμβούλιο για την Αυτάρκεια για το άρθρο 10 ε, σχετικά με την ε, συμπαραγωγή ε, είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος. Αυτό είναι το επόμενο σημείο. Μήπως μπερδέψατε τα σημεία για το 20... Όχι, όχι, για την οδηγία της ενεργειακής αποτελεσματικότητας ήθελα να μιλήσω. Κυρία Χιούμπνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ανακοίνωση συμπεριλαμβάνει ενδιαφέρουσες πληροφορίες θεμελιώδεις για το μέλλον. και αφορά στις ε, παρεμβάσεις μας ε, για να προσανατολίσουμε καλά τις νέες μας τεχνολογίες, ούτως ώστε να καταλήξουμε σε τεχνολογία με μηδενικές εκπομπές. Βέβαια σε αυτή τη φάση δεν είναι καλύτερη στιγμή για τέτοια πράγματα. Βέβαια δεν μπορούμε να το αποφύγουμε Καλό είναι να μιλάμε από τώρα για το 2050. Τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας κάτι καλό θα βγουν από όλα αυτά. Και πρέπει να το κάνουμε τώρα για να εγγυηθούμε αηφορία στις νέες γενναίες. Κάποιος από τους συναδέλφους έλεγε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές, αλλά για να το, αλλά για να το κάνουμε πρέπει να αρχίσουμε τις οικονομίες. Και θα πρέπει να δούμε προς αυτήν την κατεύθυνση, προς αυτήν την προοπτική, λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο και την οικονομική πλευρά. Πρώτα απ' όλα πρέπει να στοχεύσουμε στην οικονομία, στην ανάπτυξη οικονομίας με χαμηλές εκπομπές. Αλλά φτάνει να στοχεύουμε στην ενεργειακή αποτελεσματικότητα ή χρειάζεται και κάτι άλλο παραπάνω, δηλαδή να μπορέσουμε να επενδύσουμε στην καινοτομία, μπορούμε να επενδύσουμε στην πράσινη ενέργεια, σύμφωνοι, για να... αλλά χρειάζονται λεφτά για να γίνουν όλα αυτά και πρέπει να μπορέσουμε να στρατευτούμε σε βάθος για να πετύχουμε αυτή την καινοτομία. Χρειαζόμαστε πιο σύγχρονες μεθόδους παραγωγής για να πετύχουμε την αυτάρκεια. Πρέπει επίσης να στοχεύσουμε στην εξοικονόμηση όταν μεταφέρουμε την ενέργεια. Χρειάζονται όμως και προγράμματα για την καινοτομία, στην οικοδόμηση και κατασκευή των δημοσίων κτηρίων, των κατοικιών, των βιομηχανιών. Διότι μόνο έτσι μπορούμε να αναπτύξουμε μία οικονομία ε, με χαμηλές εκπομπές και ανάπτυξη της καινοτομίας και να μπορέσουμε δηλαδή να καταφέρουμε και κάτι έναντι των ανταγωνιστών και να βρούμε και θέσεις εργασίας. Αλλά όλα αυτά χωρίς παράδες δεν γίνονται, χωρίς χρηματοδότηση δεν γίνεται τίποτα. διότι όπως έλεγε εδώ κάποιος τέρμα με τις επιδοτήσεις δεν μπορούμε να μοιράζουμε έτσι λεφτά θα πρέπει να αρχίσουμε να δίνουμε επιδοτήσεις μόνο εκεί που αξίζει τον κόπο. Και μετά υπάρχει και κάτι το οποίο δεν μου βγει, δεν, δεν, δεν το πήρε το μάτι μου στην έκθεση. Ε, γιατί δεν μιλάμε για την ανακύκλωση και την ε, επαναχρησιμοποίηση, γιατί και έτσι εξοικονομούμε. ανακυκλώσιμα και ξαναχρησιμοποιημένα προϊόντα πάντοτε οδηγούν στην εξοικονόμηση και αποτελεσματικότητα. Κυρία Γιόρταν Σίζελη, και εγώ συμφωνώ με αυτά που λέει ο εισηγητής ότι εάν θέλουμε να ασχοληθούμε με τους στόχους για την κλιματική προστασία θα πρέπει να κοιτάξουμε τι κάνουν και οι γείτονέ μας, οι άμεσοι γείτονέ μας και οι άλλες χώρες του κόσμου. Υπάρχουν λοιπόν δύο τμήματα της προβληματικής. Από την αρχή πρέπει να δούμε τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε και μετά να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. η στόχη του 2020 είναι πραγματικά φιλόδοξη το 20% ή το 30% στη μείωση των ε, εκπομπών. Αλλά τι θα γίνει μετά από το 2020 δεν το έχουμε συζητήσει. Είναι μια πραγματική λοιπόν πρόκληση για την Επιτροπή μας και πιστεύω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε όλα αυτά τα οποία χρειάζεται ο βιομηχανικός τομέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περισσότερες επενδύσεις για το περιβάλλον και θα πρέπει να ενισχύσουμε όλες αυτές τις επενδύσεις που ανταποκρίνονται στις πολιτικές μας. Πρέπει να θέσουμε το ερώτημα αυτό. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε λοιπόν τους απαραίτητους ε, δρόμους για να προωθήσουμε αυτές πολιτικές και επέκεινα του 2020. Πρέπει να υποστηρίξουμε όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τη στρατηγική μας μέχρι το 2020, αλλά πρέπει να σκεφτούμε και για το περαιτέρω. Η Κομισιόν ζήτησε να υπάρχει μια τομεακή αντιμετώπιση για τα θέματα αυτά. Εμείς ε, φυσικά ο στόχος μας είναι να μειώσουμε τα, την εκπομπή αερίων θερμοκηπίου, αλλά συγχρόνως θα πρέπει να καθαρίσουμε μέσα εισαγωγικά και τη βιομηχανία μας, να μειώσουμε τη χρήση τεχνολογιών που εκπέμπουν αέρια του θερμοκηπίου. Και επίσης πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το θέμα της κατανάλωσης, <clears throat> του επίπεδου κατανάλωσης μέσα στην Ευρώπη. Πρέπει να εκτιμήσουμε ποιες είναι και οι εκπομπές που προκύπτουν από την ιδιωτική κατανάλωση, από την κατανάλωση των οικοκυριών στην Ευρώπη. Δεν θα έχουμε λύσει λοιπόν ποτέ πλήρως το πρόβλημα αν δεν λάβουμε και αυτό υπόψη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ζαντό, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ένας μεγάλος Ιταλός διανοούμενος που μάλλον τον ξέρετε πολύ έλεγε ότι κρίση υπάρχει όταν ο παλαιός κόσμος δεν, μπορεί να εξα... δεν θέλει να εξαφανιστεί και όταν δεν μπορεί να γεννηθεί ο νέος κόσμος. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζουμε σήμερα νομίζω στο ενεργειακό ζήτημα. Με πολύ προσοχή άκουσα τον κύριο Βιδάλ Κουάντρα, αλλά δεν είμαι σίγουρη τον κατάλαβα κιόλα ε, όταν λέει ότι δεν θέλει να υπάρχουν δημόσιε επιχορηγήσεις, επιχειρήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα κατάλαβα καλά ότι αυτό που θέλει ουσιαστικά είναι τα επιδόματα για τις ποσοστώσεις του άνθρακα επιχειρήσεις να τις καταργήσουμε, γιατί και αυτό είναι μία μορφή επιδότηση. Όταν λέει ότι πρέπει να έχουμε σαφείς φιλόδοξους στόχους σε θέματα αλλαγής του κλίματος, σωστά ερμηνεύω ότι εννοεί ότι προφανώς θα πρέπει πολιτικοί στόχοι οι ενεργειακοί, οι κλιματικοί στόχοι τους οποίους θεσπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει οι στόχοι αυτοί να ανταποκρίνονται και να αντιστοιχούν ε, στις εκθέσεις ε, και τις προειδοποίησεις των επιστημόνων. Και αν ε, είμαστε σε ένα τέτοιο σχήμα, καλύτερα θα έπρεπε σήμερα ήδη να θεσπίσουμε σημαντικούς σοβαρούς στόχους ε, από το να λέμε το 2050 θα έχουμε 95% ε, μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Ε, ας τα ξεκινήσουμε από τώρα, γιατί οι επιστήμονες αυτό μας λένε και το ίδιο θα πει και η Επιτροπή για του Κλίματος. Θα δούμε λοιπόν, ε, δεν θέλουμε να υπάρχει αστάθεια ούτε έλλειψη δυνατότητας πρόβλεψης για τις επιχειρήσεις. Αυτό θα προκύψει όμως αν δεν κάνουμε από τώρα ε, αν δεν γνωρίσουμε στόχους. Και πρέπει να σας πω ότι παρά τη Φουκουσίμα, παραδείγματο χάρη, η Ιαπωνία παραμένει στο στόχο του 25% για τη μείωση του των θερμοκηπιακών έρμων το 2020 και ε, θέλουμε ε, να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί στους στόχους μας. Άρα... Και αυτός ο στόχος του 30% δεν είναι τόσο σοβαρός όσο ο προηγούμενος που ακούστηκε. Είναι σημαντικές οικονομικές προκλήσεις. Θα πρέπει να ξαναδούμε τι σημαίνει κλιματική αλλαγή, τι σημαίνει όμως κυρίως οικονομικό δυναμικό, κοινωνικό δυναμικό μιας ενεργειακής επανάστασης. Και ένα τελευταίο σημείο, η γραμμική λίγο πολύ προσέγγιση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να είμαστε σοβαροί. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι πρέπει να γίνονται σεβαστοί οι στόχοι, άρα δηλαδή τελικά θα κάνουμε σοβαρές προσπάθειες για τιμή στον των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων. Ξέρουμε όμως, το λένε οι επιστήμονες, το λένε οι οικονομολόγοι, ότι όσο πιο νωρί στείλουμε τα σωστά ε, σημάδια και μηνύματα, λιγότερο κόστος θα προκύψει και για το περιβάλλον και οικονομικό κόστος και βιομηχανικό και κοινωνικό. Ολοκληρώνω λοιπόν. Πρέπει να έχουμε μια πολύ πιο γραμμική προσέγγιση για τις προσπάθειές μας, διότι διακυβεύονται πολλά για την επιστήμη, για τον ισότιμο ρόλο που θα παίξει ε, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του άνθρακα Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε την πρόταση της Κομισιόν, η Ευρώπη 16% θα έχει το μερίδιο με λιγότερο από 6% του πληθυσμού. Δεν είναι ανάλογα τα μεγέθη. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε τις τομές που χρειάζεται από τώρα και να μην φοβόμαστε. Ευχαριστώ. Απλώς δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Χολ, Ντέιβις, Βίδαλ Κουάδρας, και έχουμε μετά άλλα δύο σημαντικά σημεία της μέσης διάταξης. Παρακαλώ, εν συντομία. Παρακαλώ. Επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Ζαντός σε μένα, λέει ο κύριος Βιδάλ Κουάδρας, είναι θέμα καλής ανατροφής να το απαντήσω. Όχι, όχι, λέει ο πρόεδρος αν συμφωνούν όλοι να λάβετε το λόγο, εγώ δεν έχω πρόβλημα, αλλά είναι και άλλοι συνάδελφοι. Davis, Hall, Herzog θέλουν να μιλήσουν. Θέλετε να μιλήσει πριν από εσάς ο κύριος Βιδάλ Παρακαλώ, κύριε Βιδάλ Κουάδρας. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ζαντό. Όταν εγώ σας λέω ότι μακροπρόθεσμα πρέπει να εξαλειφθούν όλες οι επιδοτήσεις, δεν κάνω καμία απολύτως εξαίρεση. Όλες γιατί οι δυνάμεις της αγοράς θα πρέπει να μας δώσουν τον πιο αποτελεσματικό τρόπο να πετύχουμε τους στόχους μας, χωρίς καμία εξαίρεση. Κάτι ακόμα που θέλω να σας πω, δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ των διαφόρων στόχων της πολιτικής μας σε ό,τι αφορά τη μείωση των εκπομπών. Η μείωση των εκπομπών είναι καλή για το περιβάλλον, είναι καλή και για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας και για την ασφάλεια εφοδιασμού. Είναι ένα συνεκτικό σύνολο. Δεν υπάρχουν αντιφάσεις και τελευταίο σημείο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι βράχει πρόθεσμα η κρίση θα οδηγήσει σε σημαντικές εντάσεις για τις κυβερνήσεις τις τοπικές από αυτοδικής περιφερειακές κυβερνήσεις. Και αυτό θα έχει και αποτελέσματα στην ανεργία. Δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε αυτό. Χολ. Ευχαριστώ. Εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό να μην τα βλέπουμε όλα τα πράγματα μαύρα και σοφερά. Ο κύριος Βινταλ Κουάδρας συνήθως είναι πιο αισιόδοξο. Ίσως ε, θα μου εξηγήσει μετά γιατί δεν τα βλέπει τόσο μαύρα. Αντιμετωπίζουμε μια ρευστή κατάσταση. Πρέπει να θυμόμαστε όμως ότι αποτελεί μια απειλή, αλλά συγχρόνως και μια ευκαιρία. Μπορούμε να είμαστε πολύ πιο θετικοί για το ότι μπορούμε να προσποριστούμε από αυτές τις ευκαιρίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μας είπαν, είναι απομονωμένη. Αλλά ένας άλλος τρόπος να δούμε το θέμα αυτό είναι να δούμε ότι είναι πρωτοπόρος η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πλεονέκτημα του να είσαι πρωτοπόρος είναι ότι αν μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην οικονομία μας και στη χρήση της ενέργειας, θα αποκομίσουμε ένα μεγάλο οικονομικό <clears throat> πλεονέκτημα. Αν είμαστε οι πρωτοπόροι στην τεχνολογία χαμηλής χρήσης άνθρακος, θα είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι θα μπορούν να πουλήσουν αυτή την τεχνολογία στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν βλέπω λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι σε μειονεκτική θέση επειδή είναι μόνη της, αλλά αντίθετα να έχει πλεονεκτήματα. Δεύτερον, λέει η εκθέση του κ. Πυρίλο, ότι είναι δύσκολη η ενεργειακή αποδοτικότητα. Δεν έχουμε φτάσει βέβαια στο επίπεδο του, της μείωσης της κατανάλωσης κατά 20%. Μόνο 10% γι' αυτό έχουμε την οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Μα κάνουμε σωστά την εργασία μας και έχουμε μόλις ξεκινήσει θα είναι πολύ εύκολο για μας να φτάσουμε το στόχο της μείωσης κατά 20% στην κατανάλωση ενέργειας και αυτό θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε προς μια οικονομία χαμηλής χρήσης άνθρακα και θα κάνει το χάρτη πορείας για την χαμηλή ανθρακική οικονομία πολύ λιγότερο πολύ Όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας όταν σκεφτόμαστε αυτό το θέμα. Herzog. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λίγα σχόλια μόνο αν είμαστε τώρα πρωτοπόροι όχι. Εγώ νομίζω το θέμα είναι να έχουμε ε, το σωστό αυτό οδικό χάρτη και να τον τηρήσουμε μέχρι το 2050. Άρα ε, δεν ξέρω αν είμαστε πρωτοπόροι, αλλά πρέπει να τρέχουμε γρήγορα. Αλλιώς θα έχουμε πρόβλημα. Ε, επίσης, ο εισηγητής καταλήγει σε πολύ καλά συμπεράσματα, είναι πολύ καλή η εκθεσή του και έχω λίγες παρατηρήσεις για να είμαστε λίγο πιο συνεπείς στην παράγραφο 3 ζητά να υπάρχει μεγαλύτερη συνέπεια στα κοινωνικά, με τα κοινωνικά προγράμματα. Εγώ λέω να υπάρχει και εντό αυτών των προγραμμάτων μεγαλύτερη συνέπεια. Ιδίω όταν γίνεται λόγο για τα χρηματοοικονομικά μέσα, όπου συχνά βλέπουμε ότι δίνουμε πολλέ φορέ ε, τη ζωή μα και το αίμα μα όχι όμω τα χρήματα που απαιτούνται για διάφορα σχέδια. Και στο επόμενο πολιετέ πλαίσιο θα πρέπει να δούμε ποιε είναι οι προτεραιότητές μα για το 2050. Και πηγαίνοντας προς το 2050, έχουμε μια στάση το 2020. Πρέπει να εκπληρώσουμε πρώτα τους στόχους του 20 και μετά να πάμε μέχρι το 50. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή και είναι πολύ καλό που κάνουμε μια δήλωση για, αυτή, για τους στόχους αυτούς για το 2050. Συγχαρητήρια. Ο κύριος Ντέβις που είναι από μια άλλη επιτροπή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για την ευκαιρία να λάβω το λόγο. Είμαι ο εισηγητής για τα θέματα αυτά στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Εκτιμώ ιδιαίτερα τη συνεργασία του κύριου Λό για αυτό το θέμα. Ήθελα να μιλήσει στην Επιτροπή μας την Τρίτη. Ξεκινώντας με τη συζήτηση αυτή, είναι πιο πρασινότερη η συζήτηση στην Επιτροπή Ενέργειας από ό,τι στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Έχουν σπάσει τα στερεότυπα. Έχουμε μια πολύ σημαντική ψηφοφορία που επίκειται για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του χρόνου. Ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι ο μόνος στόχος που έχει συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρωπου είναι το 20% μέχρι το 2020 και αυτό το, αυτός ο χάρτης πορείας λέει τι πρέπει να πετύχουμε το 2050 και ενδιαμέσως το 30, 40 κτλ. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεχτεί βέβαια αυτό το χάρτη πορείας, τότε η Κομισιόν θα πρέπει να μας δώσει και τα εργαλεία για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Προς το παρόν έχει τελματώσει το θέμα αυτό στο Συμβούλιο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να αλλάξουμε τα πράγματα. Αν δεν δεχτούμε όμως αυτό τον χάρτη πορείας που έχει κολλήσει το Συμβούλιο και βρεθεί το Κοινοβούλιο να τον απορρίψει, τι μήνυμα θα δώσουμε στη βιομηχανία και στους πολίτες μας. Θα κοιτάνε οι βιομήχανοι τον αφαλό και θα αναρωτιόνται τι θα γίνει στο μέλλον. Δύο θέματα συζητήσαμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Πρώτον, πιστεύετε στην αύξηση της θερμοκρασίας. Συμφωνείτε με τους περισσότερους επιστήμονες που λέει ότι πράγματι υπάρχει ανθρωπογενής αύξηση της θερμοκρασίας και είναι επικίνδυνη. Όχι λένε ορισμένοι είναι οι ηλιακές εκρήξεις και τα ε, ηφαίστεια που δημιουργούν το πρόβλημα αυτό. Κανένα δεν το λέει στη δική σας επιτροπή. Οι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο δέχονται ότι υπάρχει ανθρωπογενής αύξηση της θερμοκρασίας. Αυτή είναι η άποψη των περισσότερων επιστήμονων. Επίσης, η Επίτροπη Περιβάλλοντος διέλαβε και το άλλο ερώτημα. Πρέπει η Ευρώπη να κινηθεί μόνη της, αν δεν υπάρχει κάποια διεθνή συμφωνία θα έπρεπε να πούμε στην Πολωνία να μειώσει τη χρήση άνθρακος για την παραγωγή ενέργειας όταν η Κίνα εξακολουθεί να φτιάνει θερμικούς σταθμούς ενέργειας. Εγώ θα επιχειρηματολογούσα, όπως είπαν και πάρα πολλοί εδώ, ότι είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης να κοιτάξει το μέλλον. Ναι, βεβαίως φτιάνει σταθμούς παραγωγής ηλεκτρισμού από άνθρακα η Κίνα, αλλά φτιάνει και σταθμούς παραγωγής που έχουν πολύ χαμηλή εκπομπή διοξιδίου του άνθρακος. Όλα αυτά προχωρούν πολύ γρήγορα. Ποιο είναι λοιπόν το μέλλον. Πιστεύουμε ότι το 2030 θα έχουμε ακόμα συμβατικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρισμού από άνθρακα. Ελπίζω ότι κανείς δεν το πιστεύει και πρέπει να δώσουμε τώρα τα σωστά μηνύματα, να, ξέρουμε, να ξέρει η βιομηχανία τι περιμένουμε από το μέλλον και να μην χάσουμε την κούρσα όπως φαίνεται ότι χάσαμε για τα φωτοβολταϊκά πάνελ προς όφελος των χωρών της από Όλα αυτά μπορούμε να τα συγκρίνουμε με την κατάσταση του Ηνωμένου Βασιλείου το 1950. Ήμασταν μια προεξάρχουσα βιομηχανική χώρα τότε. Είχαμε περάσει τον πόλεμο όμω, δεν είχαμε επενδύσει. Η Γερμανία είχε στη συνέχεια το οικονομικό τη θαύμα με τι επενδύσει, όπω και τώρα η Κίνα. Εμεί δεν έχουμε ανακτήσει τη θέση μα στο Ηνωμένο Βασίλειο, βρισκόμαστε σε μια τελμάτωση γιατί δεν δώσαμε τα σωστά μηνύματα στην, ε, ε, στη βιομηχανία. Έχουν πει πολλοί ότι μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους αυτούς στην παραγωγή ηλεκτρισμού με χαμηλή χρυσή άνθρακα. Δεν πρέπει όμως να περιορίσουμε την ε, βιομηχανία από το να χρησιμοποιήσει την πυρηνική ενέργεια ή να χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες συγκράτησης και αποθήκευσης άνθρακα όταν αυτό είναι απαραίτητο και επίσης πρέπει να διορθώσουμε και το σύστημα εμπορίας των εκπομπών γιατί αυτό οδηγεί την ε, πορεία προς χαμηλότερες εκπομπές άνθρακος. Εμείς ζητήσαμε να είναι πιο ψηλή η τιμή των εκπομπών αυτών, όχι 10 ευρώ για, την, για τον τόνο άνθρακα, διοξιδίου του άνθρακος, αλλά 30 ευρώ. Πρέπει λοιπόν να σφίξουμε λιγάκι τα λουριά, όχι το 2030 ή το 2040, τώρα, Πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις που θα πούν σε αυτούς που κάνουν τις επενδύσεις για την παραγωγή ηλεκτρισμού ότι οι επενδύσεις τους θα πρέπει να λάβουν υπόψη το τι θα γίνει στα επόμενα χρόνια γιατί ο σχεδιασμός τους είναι σε ορίζοντα 30-40 χρόνων. Αυτό θέλω να πω λοιπόν τελικά. Αλλάζει πολύ γρήγορα αυτός ο κόσμος. Όλη η οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο θα έχει μια κούρσα όπου πρέπει να είναι κάποιοι οι νικητές και κάποιοι οι, οι τιμένοι. Ας παίξουμε σωστά το το παιχνίδι για να είμαστε με, με τους νικητές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέγει ο πρόεδρος. Αν συμφωνείτε. 11 Οκτωβρίου είναι η προθεσμία για της τροπολογίας. το μεσημέρι και ερχόμαστε στο επόμενο σημείο 23 επιπτώσεις της κρίσης της χρηματοοικονομικής κρίσης στον αμυντικό τομέα. Ο κύριος Τοσενκόφσκι είναι αυτός που έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόκειται για τις ε, επιπτώσεις της κρίσης στον τομέα άμυνα στα κράτη-μέλη. Εδώ πρόκειται για μια γνωμοδότηση στην Επιτροπή προς την Επιτροπή <clears throat> Εξωτερικών Υποθέσεων. Θέλω να κάνω μονάχα μερικές ε, ε, προκατακτικές παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, ξεκινήσαμε από μία δημοσίευση για την τις επιπτώσεις της κρίσης στον αμυντικό τομέα. Αυτή η έκθεση έγινε για λογαριασμό της Επιτροπής Άμυνας και Ασφάλειας. Συζητήσαμε με διάφορους εμπειρογνώμονες και από τους εκπροσώπους των αμυντικών βιομηχανιών σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα εδώ πέρα. Η επιρροή λοιπόν της κρίσης στην, στον αμυντικό τομέα είναι ένα ζήτημα για το οποίο έχουμε πραγματικά περιορισμένη δυνατότητα να επηρεάσουμε τα πράγματα 5.000 χαρακτήρες μονάχα, 25.000 χαρακτήρες αλλά εμείς θέλουμε να έχουμε σημαντικό ρόλο στα θέματα αυτά ως Επιτροπή Βιομηχανίας. Η πρώτη παράγραφος λοιπόν της ε, εκθεσής μου λέει ότι η κρίση αυτή δεν ήταν τόσο ορατή στον αμυντικό τομέα στην πρώτη φάση όπως σε, άλλες, σε άλλους κλάδους. Αλλά υπάρχει ο φόβος ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια σειρά από καθυστερήσεις ε, στον αμυντικό τομέα και να πληγεί η ανταγωνιστικότητα και η της αμυντικής βιομηχανίας. Η δεύτερη παράγραφος αναφέρει ότι η βιομηχανία αυτή βασίζεται σε διαφοροποιημένες εθνικές πολιτικές και πρόκειται για θέματα τα οποία το κάθε κράτος τα αποφασίζει με το δικό του τρόπο. Υπάρχει απόλυτα κατακαιρματισμένο καθεστώς βιομηχανικό και διαφορετικά κριτήρια ασφάλειας και γι' αυτό είναι απαραίτητη η συνεργασία, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολη ακόμα στα κράτη-μέλη. Στο τρίτο σημείο, τονίζω ότι οι διαφορές των εθνικών πολιτικών και ιδίως ο ειδικό χαρακτήρας της αγοράς αμυντικών προϊόντων κάνει τη διαδικασία ιδιαίτερα πολύπλοκη σε όλη την Ευρώπη υπάρχει ανάγκη μεγαλύτερης συνεργασίας στον τομέα αυτό που θα παίξει σημαντικό ρόλο για να εξασφαλιστεί μια κοινή αμυντική προσέγγιση σε όλη την Ευρώπη. Ο κοινό Ευρωπαϊκό Φορέα Άμυνα παίζει ένα σημαντικό ρόλο και επίση και το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο έχει ένα ιδιαίτερο ρόλο. Τέλος, Αναφέρομαι στην τετάρτη παράγραφο στα μέσα που ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν να οδηγήσουν σε μετριασμό της χρηματοοικονομικής κρίσης και επίσης θα εντείνουν τον την συνεργασία για τα θέματα άμυνας. Είναι αυτό το νομοθετικό πακέτο του 2009. Θέλουμε εμείς να ενθαρρύνουμε την ικανότητα συνεργασίας των κρατών μελών στον τομέα αυτό, αλλά ιδιαίτερα σε αυτό τον ειδικό τομέα υπάρχουν πολλές ε, επιρροές και αλληλεπιδράσεις οι οποίες είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες και σε σημαντικό βαθμό θα παίξει ρόλο η έρευνα και η ανάπτυξη στον τομέα αυτό και ακριβώς στον τομέα αυτό είναι κεφαλαιώδης η συνεργασία των κατορμελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξασφάλιση του μέλλοντος. Επειδή δεν έχω χρόνο δεν θέλω να σταθώ σε λεπτομέρειες, απλώς θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ε, συνεργάτες μου και αυτούς οι οποίοι συνέβαλαν το έργο αυτό. Και είναι σημαντικός ο ρόλος της Επιτροπής ε, Βιομηχανίας για να έχουμε ένα κείμενο. Φυσικά η γνωμοδότησή μας έχει περιορισμένη έκταση. Απλώς θέλω να σας τονίσω ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι η 11 Οκτωβρίου για να ψηφίσουμε στις 11 Νοεμβρίου και θέλω και πάλι να ευχαριστήσω τους εισηγητές για τη βοήθειά τους και χαίρομαι για τα σχόλιά τους γιατί έχουν συμβάλει ιδιαίτερα στη βελτίωση της γρομοδότησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Οι πρώτες ιδέες που μας προτείνει Είναι καλές και πρέπει να του πω ότι ήδη υπάρχει μία έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Το λέω γιατί εγώ ήμουνα εισηγητής για την διάμεση αξιολόγηση του προγράμματος πλαίσιο. Και δεν υπήρχε Δεν υπήρχε, μάλλον εγώ πρότεινα πάντοτε η Επιτροπή μας να ασχοληθεί και με το θέμα ε, της των επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής κρίσης στον αμυντικό τομέα των κρατών, διότι η αμυντική βιομηχανία αποτελεί μία πηγή οικονομικής ανάπτυξης και πρέπει και έπρεπε, θεώρησα να το δει η Επιτροπή μας, αλλά δεν με ακούγανε μέχρι τότε. Και πιστεύω ότι πρέπει να καταλήξουμε, μας ενδιαφέρει όχι μετά από τον ψυχρό πόλεμο. Πολλά κράτη-μέλη πριν από την κρίση και όλας μείωσαν τον αμυντικό τους προϋπολογισμό. Η κρίση τι κάνει, προσθέτει ακόμη παραπάνω, έχουμε λιγότερο χρήμα δηλαδή για την παραγωγή στον αμυντικό τομέα η Μεγάλη Βρετανία με τη Γαλλία κάνανε μια διμερή συμφωνία επ' αυτού πολύ σημαντική για την έρευνα στον τομέα της άμυνας. Τα κράτη-μέλη ξοδεύουν τέσσερις φορές λιγότερο σε έρευνα στον αμυντικό τομέα από τι Ηνωμένε Πολιτείε. Νομίζω ότι πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Εμείς έχουμε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, έχουμε νομική βάση το άρθρο 45 της συνθήκης και αυτός ο οργανισμός δεν έχει κανέναν προπολογισμό στη διάθεσή του. Εμείς έχουμε την πολιτική βούληση, μπορούμε να συσπυρώσουμε πολιτικές πλειοψηφίες για να μπορέσουμε να παράγουμε αηφόρο υλικό που να χρησιμοποιείται και από την πολιτοφυλακή αλλά και από τους στρατιώτες. Η Επιτροπή μας λοιπόν συμπληρωματικά με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων θα μπορούσε να ασχοληθεί με το θέμα και να ασχοληθεί με την πτυχή ε, της έρευνας. Εγώ δεν ξέρω πρέ, κατά πόσο θα βρούμε τις πολιτικές πλειοψηφίες. Συγχαίρω τον εισηγητή. Πρέπει να βρούμε τη σωστή διατύπωση ούτως ώστε να κάνουμε οικονομίες κλίμακας από τη μια. Αλλά αν όλα τα κράτη σκεφτούν σχετικά, εμείς έχουμε ένα σωρό πράγματα εδώ, διπλωματία, ε, δασμού στα σύνορα. Ένα σωρό πράγματα μπορούμε να κάνουμε για να κάνουμε οικονομίες στα κράτη-μέλη και από επιστημονικής πλευράς να μπορέσουμε να έχουμε τους καλύτερους μηχανικούς του κόσμου, να έχουμε την καλύτερη κατάρτιση για αυτούς τους μηχανικούς. Εδώ παίζεται η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο και η αμυντική μας βιομηχανία αποτελεί Λόγω υπερηφάνειας των ευρωπαϊκών λαών, διότι η δική μας άμυνα είναι αυτή που τρέχει να υπεραμυνθεί και υπερ λαών ανά τον κόσμο. Κύριος Βίμπερ. Βέμπερ, ναι. Ο τομέας των εξοπλισμών εκπροσωπεί 240 δισεκατομμύρια ευρώ σε γύρο 4.000 άμεσες θέσεις εργασίας 1,8 εκατομμύρια ή 2 εκατομμύρια περίπου έμεσες εργασίες, 40 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές. Δεν είναι ένας παραγνωρίσιμος τομέας. Πέραν τη σημασία του σε ό,τι αφορά τη στρατηγική ανεξαρτησία και την πολιτική αυτονομία της Υπήρου μας. Όταν συρρυκνώνονται τώρα με την οικονομική κρίση οι επενδύσεις, και είναι απτό αυτό, αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα. Έχουν επιδεινωθεί τα θέματα αυτά από, την, από τον άγριο ανταγωνισμό σε διεθνές επίπεδο, ακόμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όλα αυτά θέτουν δυσκολίες στον τομέα, στον τομέα των εξοπλισμών, ακόμα περισσότερο λόγω της δυσανάλογης ισοτιμίας δολαρίου ευρώ. Λόγω της κρίσης επίσης αυξάνεται η τάση των βιομηχανών μας να βρουν την ανάπτυξη αλλού και να κάνουν στρατηγικές συμμαχίες έξω από την Ευρώπη. Αν συνεχίσει όμως μια τέτοια άποψη, τι θα γίνει με την θέλησή μας να υπάρχει μια ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη αγορά όπλων. Ο κ. Σόντι τόνισε το πρόβλημα αυτό ότι η Ευρώπη χάνει πια την τεχνολογική ικανότητα στον αμυντικό τομέα και αυτό μπορεί να γίνει κάτι το οποίο θα είναι χωρίς επιστροφή. Το 2009 οι Ηνωμένε Πολιτείε 160 δισεκατομμύρια δολάρια έδωσαν στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης μόνο 30 δισεκατομμύρια ευρώ έδειξε η Ευρώπη. Αυτό δεν θα μας επιτρέψει να παραμείνουμε στην πρωτοπορία στον αμυντικό τομέα. Δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων. Πρέπει να υπάρξει εξορθολογισμός των δαπανών, να ξεπεράσουμε τα τομεακά στεγανά και να αυξήσουμε τα κονδύλια έρευνας για να κάνουμε από κοινού όλα αυτά που μπορούμε να κάνουμε για να ευνοήσουμε μια καλύτερη σχέση μεταξύ, στρατι... μεταξύ πολιτικής και στρατιωτικής έρευνας, όπως γίνεται και σε άλλους τομείς, όπως είναι ο τομέας του διαστήματος και των τηλεπικοινωνιών. 60% από την αμυντική, παραδείγματο χάρη ε, έρευνα, έχει θετικές επιπτώσεις στην πολιτική έρευνα. Δυστυχώς, ενώ οι πολιτικοί υπεύθυνοι αυξάνουν τις δηλώσεις τους υπέρ μιας Ευρώπης της άμυνας, αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα είναι ακριβώς το αντίθετο. Τα εθνικά συμφέροντα είναι αυτά τα οποία έχουν το πάνω χέρι και η θέληση συνεργασία στον ευρωπαϊκό χώρο διαλύεται. Μετά από τα μεγάλα προγράμματα δεκαετία, δεκαετία του 1980, όπως παραγωγός χάρη το κοινό ελικόπτερο, το μεταγωγικό ε, αεροσκάφος Α400 ή το ευρωμαχητικό, κανένα πρόγραμμα δεν έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 1980 σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θέτουμε σε μεγάλη δυσκολία το σύστημα GMS για τους δορυφόρους ο καθένας προσπαθεί να διατηρήσει τις δικές του ικανότητες χωρίς να λάβει υπόψη ότι με τον τρόπο αυτό υπάρχει ο κίνδυνος να χάσουμε συνολικά τις ε, ικανότητές μας σε ένα όλο και πιο έντονο διεθνή ανταγωνισμό. Η κρίση και ο παραλογισμός της επικάλυψης σε υλικό και σε δραστηριότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να μας οδηγήσει να έχουμε καλύτερο τρόπο να αντιμετωπίσουμε τον ανταγωνισμό αυτό για να έχουμε εξοπλισμό που παράγεται πιο φθηνά και είναι καλύτερος. Χωρίς αυτή την αναδιάρθρωση θα χάσουμε και την ικανότητα ανταγωνισμού μας και την αμυντική βιομηχανία μας που θα είναι ένα φανάσιμο πλήγμα εγχειριδίου στην πλάτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει το ταχύτερο δυνατό λοιπόν να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή πολιτική η οποία θα δώσει γέννηση σε μια βάση βιομηχανική που θα ευνοεί την αμυντική βιομηχανία. Γι' αυτό ως συμπέρασμα της έκθεσης του κ. Τσερνιώσκη θέλω να υπογραμμίσω ότι οποιαδήποτε πρόοδος προς μια πολιτική άμυνας δεν πρέπει να θεωρηθεί απειλή στην κυριαρχικότητα των κρατών. Γιατί έχει τη φράση 3 η έκθεσή του Λέει ο κ. ότι μια πολιτική κοινή άμυνας είναι σημαντική από οικονομική άποψη, αλλά παρόλα αυτά κινδυνεύει να κλονίσει και να κλειδωρήσει την εθνική κυριαρχικότητα. Αν θέλει να διατηρήσει την εθνική κυριαρχία σε βάρος μιας κοινή βιομηχανίας στον αμυντικό τομέα, τότε θα χάσουμε όλοι μαζί. Πρώτα η συνεργασία και δεν μπορούμε να έχουμε όπως σήμερα όλοι διαφορετικά αμυντικά υλικά. Αλλιώς θα χάσουμε όλοι. Σας ευχαριστώ και ο εισηγητής και πάλι για να κλείσουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μόνο δύο λόγια ακόμα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που έλαβαν το λόγο στη συζήτηση αυτή και τον κύριο Όντι για την ε, απάντησή του έθεσε ένα ερώτημα. Αν τα προβλήματα αυτά θα πρέπει να τα αντιμετωπίσει η δική μας Επιτροπή. Μετά από τις συζητήσεις οι οποίες έχουν γίνει, εγώ είμαι πεπισμένος ότι αυτά τα ερωτήματα είναι δικά μας, ανήκουν στη δική μας Επιτροπή. Γιατί όλα τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την έρευνα και την ανάπτυξη είναι πολύ σημαντικά στον αμυντικό τομέα. Είναι αρρήκτο συνδεδεμένα με την βιομηχανική πολιτική. Αυτό το δείχνουν και τα γεγονότα στον περιγυρό μας, ιδίως στην Βόρεια Αφρική, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά να αναπτύξουμε τον αμυντικό τομέα. Πρέπει επίσης να σκεφτούμε ότι η υψηλή τεχνολογία αναδύεται πρώτα στον τομέα της ε, άμυνας και μετά έρχεται στον πολιτικό τομέα η Γαλλία ήταν υποδειγματική σε ό,τι αφορά την τεχνολογική ανάπτυξη που προέκυψε από την αμυντική βιομηχανία. Καταπληκτικά προϊόντα προέκυψαν από αυτή τη βιομηχανία. Γι' αυτό η Επιτροπή μας πρέπει να συζητήσει ακόμα περισσότερο και χαίρομαι για την ευκαιρία να έχουμε μια περαιτέρω συζήτηση. Ευχαριστώ. Ανέφερε ο συνάδελφος Σενόφσκι ποιες είναι οι προθεσμίες για τις τροπολογίες. Μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 24, ενεργειακή απόδοση και κατάργηση των οδηγιών 2004-8 ΕΚΡ και 2006-32 ΕΚΡ. Ο κύριος Τούρμες έχει το λόγο. Κλοντ, it's your turn. Κλοντ, εσύ είσαι. Ε, thank you, Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα λοιπόν ήθελα να σας κάνω μία εισαγωγή, να σας παρουσιάσω σε αδρές γραμμές ε, τις ιδέες μου, να ακούσω τις απαντήσεις σας και μετά κάτι που πρέπει να αποφασίσουμε είναι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Έχω στείλει στο mail σας μία πρόταση. Αρχικά είχα βάλει ως προθεσμία την 20 Οκτωβρίου, αλλά επειδή καθυστερεί λίγο η έκθεσή μου, τώρα λέω 27 Οκτωβρίου να σας προτείνω ημερομηνία. Και θα το αποφασίσουμε σήμερα. Λοιπόν, επί της ουσίας τώρα, πριν ζητήσουμε το χάρτη πορείας για το 2050, για το κλίμα δηλαδή, συζητήσαμε μετά και τη χρηματοδότηση και τον αντίκτυπο στη βιομηχανία. Είναι σαφές ότι η νομοθεσία που συζητούμε τώρα για την ενεργειακή απόδοση έχει πολύ μεγάλη σχέση αφενός με τη συζήτηση για το κλίμα και την ενέργεια, αλλά και αφετέρου με τα θέματα της χρηματοδότησης. Ένα θέμα δύσκολο φυσικά στους δύσκολους αυτούς καιρούς που ζούμε σήμερα. Όλοι όσοι εργάζονται στον τομέα του κλίματος και βλέπουν ε, τα θέματα αυτά καταλαβαίνουν ότι για να μην αυξηθεί πάνω από δύο βαθμούς η θερμοκρασία πρέπει να είμαστε πολύ φιλόδοξοι. Και στην ε, Διεθνή Επιτροπή Ενέργειας λέγεται ότι 50% και παραπάνω θα πρέπει τουλάχιστον να προέρχεται από τη βελτίωση εξοικονομήσεων στον τομέα της ενέργειας, από την ενεργειακή απόδοση. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτούς τους δύο βαθμούς. Και με την ενεργειακή απόδοση μπορούμε να μειώσουμε τις εκπομπές ε, θερμοκηπιακών αερίων με τον πιο φθηνό τρόπο. Δεύτερον, η ισορροπία των ροών της οικονομίας. Έχουμε αντιληφθεί ότι κάθε χρόνο η ευρωπαϊκή οικονομία αυτή χάνει 400 δισεκατομμύρια και παραπάνω. Ένα πλούτο που το μεταφέρουμε στους, στις χώρες που παράγουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο. 400 δις, τα οποία εκραίουν από την ευρωπαϊκή οικονομία. Είναι ο σημερινός αριθμός, το σημερινό νούμερο. Και είναι δύο παράγοντες που επηρεάζουν. Οι δικές μας πετρελαϊκές πηγές και πηγές φυσικού αέριου μειώνονται, τα αποθέματά μας, και επίσης υπάρχουν πολλές μελέτες και εμπειρογνώσια που λέει ότι επειδή οι Κινέζοι, οι Βραζιλιάνοι και άλλες οικονομίες ανθίζουν, οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου ίσως να αυξηθούν ακόμη περισσότερο από ό,τι είναι σήμερα. Αυτό που θέλω να προτείνω λοιπόν είναι ένα κούρεμα, ένα haircut στο ενεργειακό μας χρέος. Δεν θέλω η οικονομία μας κάθε χρόνο να χάνει 400 δισεκατομμύρια και ίσως και περισσότερο στο μέλλον. Με την νομοθεσία αυτή λοιπόν μιλάμε για 5 δις και κούρεμα σε αυτό το ενεργειακό χρέος. Αυτό σημαίνει 50 δις περισσότερα που θα μπορούμε να επενδύσουμε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη, στον τομέα της οικοδομής στην Ευρώπη, ενώ μπορούμε ταυτόχρονα να βοηθήσουμε και τις βιομηχανίες μας να είναι πιο παραγωγικές ενεργειακά. Και αυτό έχει σχέση και με τη σημερινή οικονομική κρίση, που είναι χρηματοπιστωτική μεν, αλλά και δημοσιονομική και κοινωνική όλο και περισσότερο. Έλεγχος του κόστους επίσης. Όταν τα δύο τρίτα της παραγωγής ισχύω θα πρέπει να καλύπτεται και ξέρουμε ότι πρέπει να αυξηθεί η τιμή του ηλεκτρισμού και αν πρέπει να εξυγχρονιστεί το δίκτυο, δηλαδή να αυξηθεί και το κόστος, δύο πτυχές ή τρεις μπορούν να βελτιωθούν με την νομοθεσία αυτή. όγκο επί τιμή, κιλοβατόρα παραδείγματο χάρη. Ε, αν αυτό είναι η τιμή, μπορούμε να παίξουμε. Ξέρουμε ότι ε, ο όγκος μειώνεται, όχι η τιμή τη κιλοβατόρα. Δεύτερον, αν είμαστε φιλόδοξοι και θέλουμε να έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας και ενεργειακή απόδοση, μπορούμε να εξοικονομήσουμε μέχρι και το 50% της απαραίτητης ε, παροχής ισχύω μέχρι το 2030. Βέβαια αυτό έχει θετικό αντίκτυπο και στο κόστος. Και η τρίτη πτυχή είναι η εξής. Στη ΣΥΠΑ δεν υπάρχει μόνο ανταγωνισμός στην αγορά ηλεκτρισμού μεταξύ των προμηθευτών, υπάρχει ανταγωνισμός και μεταξύ προμήθειας και ζήτη, προσφοράς και ζήτησης. Η οδηγία αυτή θα πρέπει να δημιουργήσει αγορά που θα ανταποκρίνεται στην υψηλή ζήτηση και θα εκεί κάποιες πιέσεις προς τα κάτω, σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή μεταξύ Παρισιού, Λονδίνου, Λιψίας και ξέρω εγώ τι σε άλλες πόλεις. Θέλουμε λοιπόν να ασκήσουμε πιέσεις προς τα κάτω. Και τέταρτο σημείο, ενεργειακή παινία. Όταν συζητάω με τους συναδέλφου μου από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, τι μου λένε, υπήρξαμε σε κομμουνιστικά συστήματα, ενέργεια ήταν τσάμπα ουσιαστικά. Και είχαμε όμως πολλούς πολίτες που έμεναν σε κτίρια που δεν είχαν καλή μόνωση. Πρέπει να έχουμε λοιπόν τη σωστή πολιτική για να μην αντιμετωπίσουμε κοινωνικές εντάσεις όπως αντιμετώπισαν πολλοί πολίτες της Ανατολικής Ευρώπης. And, uh, is το ερώτημα είναι, μπορούμε να το χρηματοδοτήσουμε και νομίζω ότι θα πρέπει. Να το σκεφτούμε γιατί έχουμε μεν εργαλεία, αλλά πρέπει να δημιουργήσουμε και άλλα. Σήμερα ο Επίτροπος Χάν θα προτείνει το 20% των, ταμείων, των, κονδύλων του Ταμείου Συνοχής να είναι για την ενέργεια και την ενεργειακή απόδοση και το 6% ...στον λιγότερο ευνοημένο περιοχών. Πολλά χρήματα που θα μπορούσαν συνέχεια να χρησιμοποιηθούν με θετικό τρόπο. Στην οδηγία αυτή επίσης, μέσω του άρθρου 6, προβλέπεται δημιουργία ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου για ε, ενεργειακές εταιρείε. Και θα πρέπει να δούμε και τις εταιρείε που εξοικονομούν ενέργεια και που μπορούν να κάνουν επενδύσεις εκ των προτέρων και να μας βοηθήσουν και εμάς με τις επενδύσεις αυτές. Τελευταίο σημείο η θέση του Συμβουλίου τα τελευταία χρόνια ήταν όχι στόχοι. Εμείς στο Κοινοβούλιο, στην έκθεση Μπένς, το Δεκεμβρίου είπαμε θέλουμε δεσμευτικούς στόχους. Τώρα η Κομισιόν μας προτείνει δεσμευτικά μέτρα. Και το Συμβούλιο ε, πλέον, οι κυβερνήσεις πλέον λένε, ε, δεν θέλουμε δεσμευτικά μέτρα. Ούτε δεσμευτικούς στόχους θέλουν, ούτε δεσμευτικά μέτρα θέλουν. Και πού μας πάει αυτό πουθενά. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση για το double track, δεσμευτική στόχη και δεσμευτικά μέτρα. Είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση με μια-δυο κυβερνήσεις που μου είπαν, τις τελευταίες μέρες έγινε αυτό, μου είπαν ότι ή τέλο πάντων είπαν ότι αρχίζουν να το σκέφτονται. Αν τα μέτρα είναι πάρα πολύ αυστηρά και παρεμβαίνουν πάρα πολύ με, το, με τις εθνικές προσπάθειες για την ενεργειακή απόδοση, ίσως ξανα... ξεκινήσει η συζήτηση για τους στόχους. Άρα πρέπει να προωθήσουμε το double track, τη διπλή αυτή διαδικασία, γιατί έτσι έχουμε περισσότερη... περισσότερα περιθώρια για να καταλήξουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για να δούμε ποιος θέλει να λάβει το λόγο. Η ο κύριο Πίπα, καταρχήν. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα στον συγητή. Κύριε Τούρμες, με ακούτε? Ποιες είναι οι οι συνέπειες που θα προκύψουν από όλα αυτά που λέτε. Είπατε στις 20 Οκτωβρίου ότι είναι πολύ νωρίς, 27 ε, Οκτωβρίου θέλετε να είναι η προθεσμία της τροπολογίας. Αυτό δεν είπατε στην αρχή. Μήπως μπορούμε να το ρυθμίσουμε μετά, λέει ο πρόεδρος. Θέλω να έχω αυτή τη διευκρίνηση για να ξέρω αν κατάλαβα καλά. Ναι, αυτό, αυτό είπε. Ναι, είναι μια πρόταση του εισηγητή βέβαια αυτό το πράγμα. Είναι μια πρόταση, αλλά θα ήθελα να αντιμετωπίσω αυτή την πρόταση γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολύ προσεκτικά αυτό το θέμα. Κύριε Τούρμες, είσαστε ένας εφάνταστος άνθρωπος, ένας δημιουργικός άνθρωπος. Ένα άτομο που είναι ευχάριστο να συζητάει κανείς μαζί του και στα θέματα της ενεργειακής ε, ε, αποδοτικότητας έχετε κάνει πάρα πολλή εργασία. Αλλά εντυπωσιάζομαι όμως από το γεγονός ότι μας παρουσιάσετε ένα τμήμα της εκθεσής σας ένα τμήμα της έκθεσης που δεν υπάρχει φυσικά ακόμα η έκθεση σε γραπτή μορφή. Είναι απλώς ένα σχέδιο εκθέσεως αυτό είναι γεγονός ότι η νομική υπηρεσία δεν έχει ακόμα αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Επίσης ότι δεν έχει ξεκινήσει καν η, η μετάφραση αυτού του κειμένου. Πώς θα μπορέσει με ένα υπεύθυνο τρόπο να μας φέρει αυτό στις 20 Οκτωβρίου να μπορέσουμε να συζητήσουμε για το θέμα αυτό και μετά να έχουμε προθεσμία τροπολογιών στις 27 Οκτωβρίου. Όλα αυτά τα βρίσκω και ανεύθυνα γιατί έχουμε τώρα μια κατάσταση η οποία θα ενδιαφέρει όλους τους συναδέλφους οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν αυτό το θέμα. Υπάρχει το θέμα της εκπροσώπησης των συμφερόντων από αυτούς που είναι στον τομέα την, της μόνωσης, των ε, ηλεκτροστροβίλων κτλ. οι οποίοι μας έχουν φέρει πάρα πολύ συγκεκριμένες προτάσεις και θέσεις. Δεν θέλω λοιπόν να γίνουν όλα αυτά υπό την πίεση ομάδων πίεσης που θέλουν να κάνει καλή δουλειά. Εγώ θα ήθελα να ακούσω και απόψεις από αυτούς που είναι από τις ε, οργανώσεις καταναλωτών, από κοινωνικές ε, οργανώσεις θα ήθελα, εφόσον ασχολούμεθα και με τις ομάδες πίεσης, να ακούσουμε όλους τους, όλες τις ομάδες πίεσης, τα εμπορικά επιμελητήρια, τα βιομηχανικά επιμελητήρια. Δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι μπορούμε να παρουσιάσουμε τώρα μια έκθεση η οποία δεν είναι ακόμα έτοιμη και μέσα σε 7 μέρες θα πρέπει να έχουμε όλοι έτοιμε έτοιμες τις τροπολογίες. Αυτό λοιπόν δεν νομίζω ότι είναι θετικό, αυτό εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα μονάχα. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε την δυνατότητα να ακουστούν και άλλες απόψεις για την αποδοτικότητα στη χρήση ενέργειας. Δεν είναι μοναχά η εξοικονόμηση ενέργειας. Θα μπορούσαμε να είμαστε λίγο πιο δημιουργικοί στον τομέα αυτό και να το δούμε το θέμα αυτό σαν παραγωγικότητα στα θέματα ενέργειας και να έχουμε μια κοινή γραμμή προς την κατεύθυνση αυτή. Σας παρακαλώ λοιπόν να καταλάβετε ότι βρισκόμαστε στην αρχή της προβληματικής ε, αυτής και γι' αυτό ήθελα να σας πω εξ αρχής ότι δεν μπορεί να σταθεί το χρονοδιάγραμμα που έχετε προτείνει. Ο Κλώτουρμες για διαδικαστικό θέμα. Το γραφείο κατάθεσης τροπολογιών έχει συμφωνήσει η έκθεση έχει περάσει από τους, από τους νομομαθείς ε, ε, μεταφραστές. Μπορεί λοιπόν να γίνει η κατάθεση τροπολογιών, λέει ο κ. Τούρμες. Δεν υπάρχει πρόσκομα με την νομική υπηρεσία. Εγώ δεν έχω κάποια επίσημη ειδοποίηση για αυτή την έκθεση, αλλά είτε πέρασε χθε το βράδυ σήμερα το πρωί, αυτό δεν έχει καμιά σημασία. Ποιο θέλει τώρα για να λάβει το λόγο. Η κυρία Ρίερα Μαδουρέλ έχει το λόγο. Από του κοιόδη συγητέ. Πρώτη κοιόδη συγητρία. Εγώ ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για την απουσία της Σαντού, της κυρίας Τόνσεν, η οποία δεν μπορεί να είναι παρούσα σήμερα και μου ζήτησε να σας παρουσιάσω σύντομα και γενικά τη θέση της ομάδας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όμως τον κύριο και να συγχαρώ τον κύριο Τούρμες για τη δουλειά του. Εγώ Η ομάδα μου πιστεύει ότι για την ενεργειακή ε, αυτάρκεια πρέπει να στείλουμε όσο το δυνατόν μεγάλη, ένα πιο έντονο μήνυμα στο Συμβούλιο. Η θέση για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα της Ευρώπης πρέπει να είναι καθαρή και εξάστερη. Θα πρέπει να έχουμε υποχρεωτικούς στόχους, με κοινή μεθοδολογία στον υπολογι... στους υπολογισμούς, όσο το δυνατόν πιο συνενετική. Πρέπει να έχουμε μηχανισμούς που θα απελευθερώσουν όλο το δυναμικό και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τους ε, μηχανισμούς ε, για την ενεργειακή απόδοση, απόδοση και όπου θα συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αναβληθεί για αύριο. Αυτοί οι οποίοι σήμερα θα προχωρήσουν στην ενεργειακή απόδοση θα έχουν ωφέλη αύριο Γι' αυτό και είναι κατεπήγον να λάβουμε την απόφαση τώρα και να ξεκινήσουμε όσο το δυνατόν νωρίτερα. Αυτοί οι οποίοι θα έχουν αυτάρκεια στην ενέργεια μέσα στην κρίση θα είναι αυτοί οι οποίοι θα μπορέσουν να αντισταθούν παγκοσμίω, θα έχουν θέσεις εργασίας, θα μπορέσουν να διασφαλίσουν θέσεις εργασίας και επενδύσεις. Γι' αυτό κύριε η ομάδα μου θα ήθελε να είναι όσο το δυνατόν πιο βράχοι πρόθεσμες οι προθεσμίες και για την κατάθεση τροπολογιών. Αν εσείς θέλετε να το διευρύνουμε από 25 στα 27 θα το δεχτούμε, όχι όμως παραπάνω. Για όλους τους λόγους που ανέφερα. Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν ανεύθυνο να, διε... να... να μακρύνουμε την προθεσμία ε, ε, περισσότερο. Ε, ο κλάδος θα μας ευχαριστήσει διότι θέλει να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα, πιο γρήγορα και οι και όλοι οι συζητητές και όλοι οι συνεργάτες είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε όσες ώρες χρειάζεστε για να τελειώνουμε πιο γρήγορα. Εμείς εργαζόμαστε για τη δική μας ασφάλεια. Μείωση της κατανάλωσης σημαίνει ενίσχυση της αυτάρκειας. Επίσης θέλουμε να μειώσουμε την οικολογική τις οικολογικές επιπτώσεις. Κανένας δεν αμφιβάλλει για την αηφορία των, οικονομικών, των οικονομιών μας μακροπρόθεσμα. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να λύσουμε το πρόβλημα. Είναι πραγματικά μεγάλη ευχαρίστηση το να εκφράζει κανείς τη γνώμη της κυρίας Μπρίτα Τόμσον για να προχωρήσουμε προς μια αποτελεσματική οδηγία για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα που να εγκριθεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Ευχαριστώ. Πάλι μια παρατήρηση σε διαδικαστικό επίπεδο. Η ιδέα ήταν να συζητήσουμε σήμερα την έκθεση και κανονικά θα πρέπει να είναι η μετάφραση του κειμένου διαθέσιμη, που φυσικά δεν είναι διαθέσιμη. Παρ' όλα αυτά θέσαμε το θέμα στην ημέρησια διάταξη, γιατί θέλαμε να κερδίσουμε χρόνο. Πρόκειται τώρα για την πρώτη φυσικά συζήτηση, η οποία γίνεται χωρίς το κείμενο. <clears throat> Στις 20 Οκτωβρίου θα είναι η πρώτη ευκαιρία που θα έχουμε το κείμενο με τη μετάφραση και στη συνέχεια θα συζητήσουμε τις περαιτέρω προθεσμίες. Θέλω να ζητήσω από όλες τις πολιτικές ομάδες να συζητήσουν και να βρουν σε μια συνένεση ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην εκπόνηση αυτής της έκθεσης. Είχαμε περάσει κάποια στιγμή πριν από μερικά χρόνια ένα πακέτο που αφορούσε θέματα παγκοσμιοποίηση με υπερβολική ταχύτητα. Και γι' αυτό εγώ προσωπικά έχω αναλάβει το, την υποχρέωση να εξασφαλίσω ότι όλοι οι συνάδελφοι, όχι μόνο ο εισηγητή και οι σκηνιώδει εισηγητέ, όχι μόνο οι συντονιστέ και οι πρόεδροι, όλοι να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν πλήρω στην επεξεργασία μια έκθεση. Γι' αυτό σα λέω και πάλι θα προσπαθήσω όλοι οι συνάδελφοι να έχουν τα ίδια καθήκοντα και τα ίδια δικαιώματα να προσκαλέσουν εμπειρογνώμονες για ακροάσεις και τα λοιπά. Και κάπως ενοχλούμε ότι κανένας δεν ρώτησε τον πρόεδρο για, την, ε, ε για τα σχέδια του, του χρονοδιαγράμματος. Ο κύριος Τούρμες δεν με ρώτησε καθόλου για αυτές τις ε, προθεσμίες, ούτε και για τα εργαστήρια τα οποία έχουν προταθεί να γίνουν. Θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω να σκεφτείτε με λογικό τρόπο ποιο είναι ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο μπορεί να σταθεί. Σας είπα, συζητάμε πρώτα σήμερα παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμιά έκθεση. Είναι δεδομένο επίσης ότι στις 20 θα συζητήσουμε όταν υπάρχει το κείμενο και τότε μονάχα θα πρέπει να συζητήσουμε για τις περαιτέρω προθεσμίες. Υπάρχουν πολλοί που θέλουν να λάβουν το λόγο. Ο κύριος Ρόλ έχει το λόγο. Κυρία Χόλ, συγγνώμη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να επανέλθουμε εκεί που αρχίσαμε με την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση, δηλαδή τις πολιτικές δεσμεύσεις του 2007. Οι στόχοι 20-20-20 δηλαδή. Και τι τελικά είναι η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση, ουσιαστικά λέει πώς θα πετύχουμε αυτούς τους στόχους. πρέπει αυτό το έχουμε υπόψη μας όταν συζητούμε για τις εξοικονομήσεις και πώς τις ορίζουμε, γιατί θα πρέπει να είναι εξοικονομήσεις. Οικονομίες χρειαζόμαστε αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε την ενεργειακή απόδοση και τις εξοικονομήσεις τις σχετικές στο 2020. Είναι πλαίσιο, στο πλαίσιο αυτού του πακέτου. Έχουμε την αλλαγή του κλίματος, αλλά δεν είναι ο μόνος λόγος. Ε, και σε σχέση και με την κρίση που βιώνουμε σήμερα πρέπει να έχουμε μια απόλυτη μείωση σε ό,τι αφορά και την ενεργειακή ασφάλεια, ο μίλητρια, και στο πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οικονομικά ε, την ενέργεια για να είναι πιο ανταγωνιστικές οι επιχειρήσεις μας. Η Κομισιόν με την οδηγία αυτή προτείνει συγκεκριμένα μέτρα και όπως προαναφέρθηκε τα κράτη-μέλη κάπως αμφιταλαντεύονταν και άλλαξαν απόψεις για το τι θέλουν από την Κομισιόν. Και από τις δικές μου συνομιλίες και επαφές κατάλαβα ότι απέναντι σε συγκεκριμένα μέτρα τα οποία προτείνει η Κομισιόν και τα οποία δεν φαίνεται να εντάσσονται και πάρα πολύ ομαλά ε, σε κάποια πράγματα που κάνουν ήδη τα κράτη-μέλη. Κάποια κράτη-μέλη λοιπόν διερωτώνται πέραν σε αυτά τα μέτρα μήπως θα ήταν καλύτερα αν είχαν εθνικό στόχο και εκεί θα μπορούσαν με μεγαλύτερη ευελιξία να προσπαθήσουν να τον πετύχουν. Εγώ υποστηρίζω την διπλή αυτή προσέγγιση, το two-track approach, γιατί θα μας δώσει μια ευελιξία για να μπορέσουμε κάποιες από τις ανησυχίες αυτές ε, χωρών που κάνουν πολλά για την ενεργειακή απόδοση ήδη να τις καθησυχάσουμε. Μπορεί βέβαια αυτά που κάνουν να μην ε, τηρούν απόλυτα αυτά που προτείνει η Κομισιόν με την πιο αυστηρή λεπτομέρεια. Θα ήθελα τώρα να αναφέρω δύο συγκεκριμένου τομεί. Ο πρώτος είναι τα κτίρια. Στο άρθρο 6 εισάγεται η ιδέα ότι θα πρέπει το 3% των δημόσιων κτηρίων κάθε χρόνο να ανακαινίζονται. Με τα εφιστάμενα κτίρια σίγουρα έχουμε πρόβλημα. Το ξέραμε. Και τότε που ε, δημοσιεύτηκε η οδηγία για την ελληνική απόδοση των κτίριων, το 78% των κτίριων που υπάρχουν σήμερα θα, θα υπάρχουν και το 2050. Αν, κάνουμε, λοιπόν, αν δεν κάνουμε τίποτα με τα κτίρια, δεν πρόκειται να πετύχουμε εξοικονόμηση ενέργειας από τα κτίρια, τουλάχιστον στον βαθμό που χρειαζόμαστε τη μείωση. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη με τον τρόπο τους, να μην τους επιβάλλουμε εμείς, αλλά να τα πείσουμε να έχουν έναν οδικό χάρτη μέχρι το 2050 για το πώς θα αντιμετωπίσουν ε, το θέμα με τα κτίρια. Και αυτή η πρόταση της Κομισιόν, το 3%, καλοδεχούμενη είναι, γιατί κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Ο δημόσιος τομέας πρέπει κάτι να κάνει για να αναπτύξει ε, την ε, ικανότητα και της, αγοράς ε, να δώσει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, δυνατότητα επιταχύων και να μπορέσουν να κάνουν αυτές τις ανακαινήσεις. Αλλά είναι λίγο περιοριστικός ε, ο τρόπος που κάνει αυτές τις προτάσεις η Κομισιόν. Επί της ουσίας όμως το να δούμε τις ανακαινήσεις και να τον ισχύει αυτό το δημόσιο αυτό είναι, είμαι υπέρ. Δεύτερον, υποχρέωση εξοικονόμηση ενέργειας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί πετυχαίνουμε κάτι, 1,5% το χρόνο. Κάποια κράτη-μέλη έχουν ήδη υποχρέωση εξοικονόμηση ενέργεια, κάποια όχι. Αλλά όποιο κράτο μέλο έχει αυτό το στόχο, ε, βλέπουμε ότι εκεί είχαμε αποτελέσματα. Και είναι καλό να υπάρχει η ευρωπαϊκή νομοθεσία αυτή, αλλά βέβαια πρέπει να διδαχθούμε και από τι βέλτιστε πρακτικέ. Έχουμε ένα μηχανισμό εδώ που λειτουργεί, που αποδίδει, άρα είναι πολύ σημαντικό να τον αξιοποιήσουμε είναι κάτι που μπορούμε να το εμπιστευτούμε. Και ίσως χρειαστεί ευελιξία σε σχέση με τη διατύπωση. Αλλά η αρχή νομίζω ότι είναι κάτι που μπορούμε να εμπιστευτούμε, ότι μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα με αυτή την οδηγία και κάτι που έχουμε δεσμευτεί να πράξουμε το 2007. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, μια τελευταία λέξη. Δεν κατάλαβα τώρα ε, ποια είναι η διαφορά μεταξύ μου και του κυρίου Πίπερ. Εγώ πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά τα άτομα που λέει ήρθαν και σε μένα, ε, σε Business Europe ε, και πολλοί από όλα τα κομμάτια της βιομηχανίας, ΜΚΟ. Ε, ουσιαστικά μου είπαν τα ίδια που συζητούνται τόσο καιρό. Ο διάλογος έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό, δεν είναι κάτι καινούριο. Εμένα δεν, δεν μου δημιουργεί κανένα πρόβλημα η 27 Οκτωβρίου που προτείνεται ω ημερομηνία για την κατάθεση των τροπολογιών. Ήδη δουλεύουμε πάνω στο θέμα εδώ και κάποιο καιρό και νομίζω ότι θα έχουμε χρόνο για να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Ευχαριστώ. Η κυρία Φόρντ. Ευχαριστώ πολύ. Όταν εγώ δέχτηκα να είμαι σκιώδης εισηγήτρια θεώρησα ότι θα ήταν ένα εύκολο, όχι αμφιλεγόμενο και απλό θέμα. Μεγαλύτερη αποδοτικότητα, εξοικονόμηση για τις επιχειρήσεις, μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να μειώσουν το κόστος θέρμανσης και των σπιτιών τους. Το θέμα όμως αυτό γίνεται ιδιαίτερα επίμαχο και ιδιαίτερα ε, δυνητικά πολυδάπανο και διευθυντικό νομοθέτημα. Δεν θα, μια, νομοθετική, μια διευθυντική έκθεση. Δεν θέλω να πάνε τα πράγματα έτσι. Η ενεργειακή αποδόση θα πρέπει να είναι ένας, ένα μέσο να βοηθήσουμε τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις να εξοικονομήσουν χρήματα και να μας βοηθήσουν να επανέλθουμε σε οικονομική ανάπτυξη. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, εγώ προσωπικά μπορώ να έχω τροπολογίες μέχρι τις 27 του μηνός. Αλλά αυτό επειδή παρακολουθώ αυτό το θέμα εδώ και πολλούς μήνες και είχα το κείμενο αυτό στα αγγλικά που είναι στη γλώσσα μου. Αλλά αν όλα τα μέλη από τις διάφορες χώρες θέλουν και πρέπει να συμμετάσχουν σε, σε αυτή την έκθεση με τρόπο που να μην είναι αμφιλεγόμενος, θα πρέπει να έχουν όλοι το χρόνο να δουν τις τροπολογίες. Δεν μπορώ να τονίσω αρκετά πόσο σημαντικό είναι το μέτρο αυτό για να τονώσουμε την οικονομική ανάπτυξη, αν βρούμε τη σωστή λύση. Γι' αυτό θέλω να παρακαλέσω και τον Πρόεδρο να δει αν μπορεί να βρει να γίνει μια πιο ε, έγκαιρη συνεργασία του Κοινοβουλίου με το Συμβούλιο. Δηλαδή, να μην περιμένουμε μόνο την Ολομέλη για να αρχίσουμε συζητήσεις με το Συμβούλιο και την Κομισιόν, <clears throat> να μην περιμένουμε μονάχα την τυπική διαδικασία, να προχωρήσουμε πιο γρήγορα και θέλω να σας ενθαρρύνω να εξασφαλίσετε ότι δεν θα μπλοκαριστούμε μεταξύ ημών και της Επιτροπής Περιβάλλοντος για τα θέματα αυτά. Θα πρέπει όλοι να προσπαθήσουν <clears throat> να προχωρήσουν με το ταχύτερο δυνατό ε, χρονοδιάγραμμα. Είπαν ορισμένοι ότι ο τρι, τριγωνικός διάλογος δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο τον επόμενο Μάιο ή τον επόμενο Ιούλιο. Α χρησιμοποιήσουμε σωστά λοιπόν το χρονοδιάγραμμα. Για να κάνουμε αυτούς που εκπροσωπούμε του εκλογείς μας να δουν τα πλεονεκτήματα αυτής της ρύθμισης, Θέλουμε να του τονίσουμε ότι όταν μιλάμε για ενεργειακή απόδοση μας ενδιαφέρει η σχέση κόστους-οφέλους. Και αυτό είναι αυτό που προσπάθησαν να κάνουν πολλές χώρες και στα σπίτια, στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. <clears throat> Αν ζητάμε λοιπόν από τους καταναλωτές να πληρώσουν για βελτίωση στα σπίτια τους, θα πρέπει να δούνε και οικονομικό όφελος το οποίο θα προκύψει από την ανακαίνιση των σπιτιών τους. Φοβάμαι ότι σε ορισμένα κράτη οι καταναλωτές έχουν δει υψηλότερα τιμολόγια ενέργειας, αλλά δεν έχουν δει καμιά εξοικονόμηση δεν είχα ακόμα τη δυνατότητα να δω το οικονομικό τμήμα που έχει προσθέσει ο εισηγητής, αλλά το να δώσουμε στα κράτη-μέλη ένα μενού από το οποίο μπορούν να επιλέξουν ποια μέτρα θέλουν για να βοηθήσουν τον κόσμο να επενδύσει σε καλύτερες ε, ε, πρακτικές, αυτό είναι καλύτερο από το να έχουμε ένα μονάχα κατάλογο μέτρων. μέτρων. Υπάρχουν ορισμένα αμφιλεγόμενα σημεία εδώ. Το άρθρο 4 για τις δημόσιες αρχές και τα δημόσια κτίρια. <clears throat> Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα το οποίο παρακολούθησε όταν ήρθα στο Κοινοβούλιο. Η οδηγία για την ενέργεια και την εξοικονόμηση. Πρέπει όμως να έχουμε υπόψη μας ότι σε διάφορα κράτη-μέλη υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα τοπικών κυβερνήσεων, διαφορετικοί φορείς οι οποίοι στεγάζονται σε δημόσια κτίρια και η εφαρμογή αυτού του μέτρου θα μπορούσε να είναι πολύ πεπλεγμένη. Νομίζω ότι κάθε επίπεδο τοπικής, περιφερειακής, κεντρικής κυβέρνησης θέλει να εξοικονομήσει χρήματα και η ενέργεια, η εξοικονόμηση ενέργειας είναι τρόπος για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Αλλά η τωρινή διατύπωση του κειμένου, αν έχουμε μια αρχή η οποία έχει ήδη εκπληρώσει τα 99% του των απαιτήσεων για οικονομική εξοικονόμηση, θα έπρεπε και πάλι να εργαστεί για το τελευταίο 1%. Δεν έχει νόημα αυτό. Θα πρέπει να επιτύχουμε τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα με καλή σχέση ωφέλεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το άρθρο 6 για την εξοικονόμηση 1,5% ακόμα και οι χώρες οι οποίοι που έχουν συστήματα και τα οποία δεν μπορούν από τις υποχρεώσεις που έχουν για μετασκευή κτηρίων να καλύψουν το 1,5% τουλάχιστον θα πρέπει να έχουν μια επιλογή άλλων μέτρων για να μπορέσουν να επιτύχουν το στόχο του 1,5%. Εμένα δεν μου αρέσει το γεγονός ότι επιβάλλεται το 1,5% σε αιτήσια βάση. Πολλές φορές για να λειτουργήσουν αυτά τα συστήματα χρειάζεται πολλή εκπαίδευση και κατάρτιση, δημιουργία ειδικοτήτων και προσόντων. Θα πρέπει να επιτρέψουμε λοιπόν στα κράτη να τα κάνουν αυτά με το δικό τους ρυθμό ώστε να λειτουργήσουν πρακτικά και λογικά. Και φυσικά ο κύριος γνώμονας θα πρέπει να είναι η σχέση κόστους-οφέλους. Για το άρθρο 7, για τον έλεγχο και την παρακολούθηση, δεν θέλουμε εδώ πέρα να αυξήσουμε το χαρτοβασίλειο και τη γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις. Ο πρώτος έλεγχος νομίζω ότι είναι αυτός ο οποίος σημαντικός για την ευφυά τιμολόγηση υπάρχει ένα σημείο πέρα του οποίου δεν είναι πια ε, σωστή σχέση κόστους ωφέλους στην ευφυά τιμολόγηση. Δεν υπάρχει λοιπόν ε, επαρκής <clears throat> λύση με την ευφυά τιμολόγηση. Πρέπει να έχουμε και ευφυέστερες συσκευές. Το άρθρο 10 για την συμπαραγωγή. Πήγα την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα καταπληκτικό εργοστάσιο στο δικό μου ε, στη δική μου εκλογική περιφέρεια συμπαραγωγή θερμότητος και ηλεκτρισμού, είναι φανερό ότι είναι πολύ πιο αποτελεσματικό να παράγει κανείς πρώτα τον ηλεκτρισμό και μετά την ε, θερμότητα. Η θερμότητα είναι πολύ πιο δύσκολη βέβαια από τον ηλεκτρισμό να διανέμεται. Ο τρόπος με τον οποίο έχει διατυπωθεί αυτό από την Κομισιόν είναι πάρα πολύ υπαγορευτικού χαρακτήρα και περιοριστικό Πρέπει να ενθαρρύνουμε τη συμπαραγωγή όπου είναι ε, πρόσφορη και δίνει κάποια αποτελέσματα, αλλά τελικά θέλουμε να κάνουμε και εξοικονόμηση κόστους και μείωση διοξιδίου του άνθρακος. Αλλά το άρθρο αυτό θα πρέπει να είναι ε, ένα άρθρο που δεν περιλαμβάνει και την πυρηνική ενέργεια. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις χώρες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν την πυρηνική ενέργεια να τονίσουμε πρώτα την καλή χρήση της θερμότητος και όχι μοναχά την καλή χρήση του ηλεκτρισμού. Είναι σημαντικός ο τρόπος με τον οποίο το λέμε. Αν εγώ έκανα τις διαπραγματεύσεις αυτές με το Συμβούλιο, θα ήθελα προηγουμένως να υπάρχει συνένεση μεταξύ του Κοινοβουλίου και των κρατών μελών και όχι απλώς μία σύγκρουση. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε, θέλουμε συνένεση Κοινοβουλίου και κρατών μελών για τα θεμελιώδη θέματα και ιδίω συνένεση και με τους πολίτες μας που αυτούς θέλουμε να βοηθήσουμε. Εντάξει, ακούσαμε τους ε, εισηγητέ. Ίσως την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να προσπαθήσετε να είστε πιο σύντομοι. Ευχαριστώ. Όπως ε, και με το προηγούμενο έγγραφο για τους μελλοντικούς στόχους με το 2050 ασχολούμαθα με ένα θέμα πολύ συγκεκριμένο, ενεργειακή αυτάρκεια και κατάργηση οδηγών. Από όσα πληροφορήθηκα δύσκολα μπορούμε να αυξήσουμε την ενεργειακή απόδοση μέχρι το 20% το 2020. Προς στιγμή μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα εμπόδια για την προσέγγιση του στόχου, αλλά φαίνεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολο αυτό. Όλοι λένε ότι πρέπει να αυξήσουμε τις επενδύσεις για τη βιομηχανία, μετά έχουμε και τις περιφέρειες που ζητούν χρήμα για την εξοικονόμηση ενέργειας και κατά συνέπεια την αύξηση της αποτελεσματικότητας χρησιμοποιώντας νέες μεθόδους, καλύτερη μόνωση των κατοικιών κλπ. Για την οικιακή κατανάλωση και εδώ απαιτούνται επενδύσεις που θα μας επιτρέψουν να μειώσουμε με την εξοικονόμηση ενέργεια. Αλλά θα κάνουμε όλα αυτά, τι πετυχαίνουμε, διότι η ενεργειακή αποτελεσματικότητα και απόδοση σωστή σημαίνει τι σημαίνει κέρδος και ωφέλεια για την κοινωνία. Αν έχουμε μία μεγαλύτερη ενεργειακή αποτελεσματικότητα, θα μπορέ, δηλαδή θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο τη βιομάζα αξιοποιώντας τα απόβλητα της γεωργίας. Ε, πρέπει να τα δούμε όλα αυτά υπό την οπτική του κέρδους. Πρέπει να εξηγήσουμε στους πολίτες πόσα λεφτά θα κάνει την οικονομία στο λογαριασμό της ΔΕΗ άμα έχετε καλύτερα μονομένα σπίτια. Και πιο πρέπει να επιμείνουμε στο κόστος και στα πλεονεκτήματα έναντι των πολιτών. Αυτή θα, αυτό θα είναι και το πρώτο κοινωνικό κέρδος. Οι πολίτες θα ξέρουν ότι η εξοικονόμηση ενέργεια σημαίνει κερδίζω απαλού. Αυτό είναι ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Και οι αρχιτέκτονες μηχανικοί θα πρέπει να φτιάχνουν πλέον μονομένα κτίρια. Αυτό είναι αποτελεσματικότητα. Ο κ. Ζάμστοκ που είναι σχεδόν συγητής, τον οποίο τον ξέχασα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τρεις σύντομες παρατηρήσεις σε αυτή τη σημαντική πρόταση. Η ενεργειακή απόδοση δεν είναι το ίδιο με την εξοικονόμηση ενέργειας και δεν είναι ξεκάθαρη διάκριση αυτή στην έκθεση. Πρέπει να το συζητήσουμε πιο προσεκτικά αυτό το θέμα, γιατί η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να γίνει το αντίθετο, να, ε, έχει, να πάει προς την αντίθετη κατεύθυνση αν δεν το αντιμετωπίσουμε με το σωστό τρόπο. Δεύτερον, στόχοι, το 1,5% της μείωσης, συμπαραγωγή υποχρεωτική δεν είναι εύκολα εφικτά από τεχνικής πλευράς. Για πολλά κράτη-μέλη αυτό θα σημάνει πολύ μεγάλες δυσκολίες. Τρίτη παρατήρηση. Το όλο πλαίσιο πολύ λίγο συνάδει με την οικονομία της αγοράς. Παραλαμβάνω δεν είναι συμβατό με την οικονομία της αγοράς. Είναι πιο πολύ σαν ένα σύστημα διανομής. Question is if I am sitting in industrial and research and Σαν τα συστήματα που μεράζουμε σε περίπτωση πολέμου. Okay. And Axel brothers. Ο κύριος Φάνκος. Merci monsieur le président, mille excuses encore d'avoir anticipé. Χαριστόπολη. Θα είμαι πολύ σύντομο, συγγνώμη που πήρα το λόγο πιο γρήγορα από όσο έπρεπε. Λοιπόν, όπω ε, είπαν και οι συνάδελφοι, ε, είναι εξαιρετική βάση για τη συζήτηση το έγγραφο αυτό, αλλά σίγουρα χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για να μπορέσουμε να εμπλουτίσουμε το κείμενο και να το προσαρμόσουμε. Και ακούσαμε τι είπε και η σκιώδηση συγγήτρια, ότι δηλαδή το σημαντικό είναι όχι να υπαγορεύουμε, αλλά να πείθουμε. Ούτε μπορούμε να βάλουμε πάρα πολύ ψηλά τον πύχη σε χώρες που δεν μπορούν να πετύχουν τους στόχους. Αυτό θα είναι συνώνυμο της αποτυχίας. Άρθρο 10. Συμπαραγωγή ενέργειας. Ένα πολύ συγκεκριμένο άρθρο, ίσως υπερβολικά ε, συγκεκριμένο. Εγώ από την δική μου πλευρά θα έλεγα ότι καλό είναι να είμαστε πιο ευέλικτοι ώστε τα κράτη-μέλη να έχουν την επιλογή να επιλέξουν το ενεργειακό μείγμα που τους βολεύει σύμφωνα και με το άρθρο 194 της συνθήκης. Να μην επιβάλλουμε στα κράτη-μέλη την επιλογή της συμπαραγωγής. Στο σημείο 3, στο ίδιο άρθρο, η οδηγία επιβάλλει ότι οι νέες εγκαταστάσεις ε, θερμικής παραγωγής ενέργειας ε, όταν ε, πάνω από 20 ΜΒ είναι η δυνατότητα θα πρέπει να έχουν και δυνατότητα συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης θα πρέπει να έχουμε και οικονομικά και τεχνικά κριτήρια πολύ συγκεκριμένα. Επίσης γίνεται λόγος ε, για υψηλή απόδοσης εγκαταστάσει. Τι θα γίνει όμω με τις μικρούς απόδοση εγκαταστάσει τα σχέδια μικροπαραγωγής δεν θα πρέπει ε, να πνιγούν όταν θέλουμε να κάνουμε μεγάλες εξοικονομήσεις στην ενέργεια. Λοιπόν, θα κάνω κάποιες τροπολογίες και σε ό,τι αφορά αυτές τις εγκαταστάσεις μικρής δυναμικότητας, μικρής απόδοσης. Και θα ήθελα να επιμείνω επίσης και στη σημασία γενίκευση των εγκαταστάσεων συμπαραγωγής ε, με βάση τα απόβλητα και νομίζω ότι θα πρέπει να το ε, εξετάσουμε εκ νέου και υπό το πρίσμα των νέων οικονομικών εργαλείων. Ευχαριστώ. Κουάδρας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. και εγώ θέλω να χαιρετήσω καταρχήν αυτήν την τόσο αναμενόμενη πρόταση της Κομισιόν. Είμαι πεπισμένος ότι είναι καιρός η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεκινήσει τις επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση με ένα ευφυή και ανταγωνιστικό τρόπο. Το να ορίσουμε τι σημαίνει ευφυής και ανταγωνιστική ενέργεια είναι ακριβώς ο στόχος και το καθήκον και η πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει η Επιτροπή μας. Λίγα σχόλια μονάχα σε σχέση με ορισμένα σημεία όπου έχω ανησυχίες γιατί αυτά τα οποία με τα οποία συμφωνώ δεν χρειάζεται να τα θίξω. Θέλω καταρχήν να εκφράσω τις αμφιβολίες μου για τη μέθοδο που προτείνεται από την Κομισιόν για την καταμέτρηση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Αφορά μονάχα την πρωτογενή κατανάλωση. Αλλά εγώ θεωρώ ότι το να τεθούν ανώτατα όρια δεν είναι ο τρόπος να μειώσουμε την ενεργειακή κατανάλωση. Μία σωστή παράμετρος είναι η ένταση εργασίας. Η ενέργεια λοιπόν που καταναλώνεται ανά μονάδα ΑΕΠ. Αυτός πρέπει να είναι ο τρόπος με τον οποίο θα καταμετρούμε την ε, ενεργειακή αποδοτικότητα. Αυτό γίνεται και από τους οικονομολόγους της ε, αναδυόμενες οικονομίες. Δεύτερον, οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις εταιρείες παραγωγής ενέργειας από το άρθρο 6. Ειλικρινά δεν θεωρώ ότι το να υποχρεώσουμε τις εταιρείες να μειώσουν τις πωλήσει ενέργειας ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει μια λύση. Είναι καλύτερα να έχουμε φορολογικά κίνητρα. Οι επιδοτήσεις για την ε, εξοικονόμηση. Τίποτα όμως από όλα αυτά δεν βρίσκεται στην πρόταση της Κομισιόν. Χρειαζόμαστε μηχανισμούς ανάκτησης του κόστους από τις επιχειρήσεις αν τους επιβάλλουμε πρόσθετο άχθος υποχρεώσεων. Επίσης, το τρίτο σημείο αφορά τα άρθρα 4 και 5 τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στα δημόσια σώματα για τα κτίρια και την επισκευή, η ανακαίνιση ή αγορά νέων κτίριων. Το να κάνουμε τα δημόσια, τις δημόσιες αρχές ως την, τον κύριο Μοχλό να προωθήσουμε νέες υπηρεσίες στον τομέα της ενέργειας, αυτό είναι θετικό. Αλλά φοβάμαι ότι τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο οι δημόσιες περιφερειακές και τοπικές αρχές δεν θα μπορέσουν να το επιτύχουν αυτό γιατί υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη λιτότητος. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές σε σχέση με τη δυνατότητα όλων αυτών των δημοσίων φορέων να επενδύσουν στην εξοικονόμηση ενέργειας όσο ε, συνεχίζεται η οικονομική κρίση. Κάποια ακόμα σχόλια σε σχέση με την πρόταση να προωθήσουμε τη συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού. Εγώ πάντα έχω υποστήριξει την αρχή της συμπαραγωγής και έχω τον Όρμπερτ Γκλάντε μπροστά μου που έχουμε συνεργαστεί μαζί του και έχουμε καταφέρει να περάσουμε ε, πάρα πολλά πράγματα στην πρώτη οδηγία για την συμπαραγωγή. Είμαι πεπισμένος ότι η συμπαραγωγή είναι κάτι το οποίο μπορεί να βελτιωθεί ακόμα στο μέλλον. Επομένως χαίρομαι για την ιδέα αυτή της συμπαραγωγής, αλλά πρέπει να είμαστε, ε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Γιατί δεν μπορεί να λάβουμε μονάχα την ε, συνολική παραγωγή σαν κριτήριο για τη συμπαραγωγή. Πρέπει να λάβουμε υπόψη το δίκτυο διανομής τα τις, τα σημεία συμφόρησης στο δίκτυο διανομής. Δεν μπορεί λοιπόν μονάχα το επίπεδο θερμότητας που παράγεται να είναι το μόνο κριτήριο. Χρειαζόμαστε μια συνολικότερη προσέγγιση. Ας επιβάλλουμε την συμπαραγωγή όταν όλοι οι απαραίτητοι παράγοντες ε, έχουν εξασφαλιστεί και όχι μονάχα η ζήτηση για θερμότητα. Όταν λειτουργεί λοιπόν και το δίκτυο με τον κατάλληλο τρόπο. Ένα τελευταίο σχόλιο για το χρονοδιάγραμμα. Ειλικρινά. Πιστεύω ότι μια οδηγία τέτοιας σημασίας και τέτοιας φιλοδοξίας που έχει τεράστιες συνέπειες για την οικονομία μας. Θα πρέπει να μελετηθεί και να τύχει επεξεργασίες από την Επιτροπή μας μέσα σε ένα επαρκές χρονικό διάστημα. Παρακαλώ λοιπόν να μην έχουμε βεβιασμένες κινήσεις και ας δώσουμε σε όλους τους συναδέλφους τη δυνατότητα να συμβάλλουν στην εκπόνηση αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Φόρτια, διαδικαστικό θέμα. Ευχαριστώ. Ίσως έχετε δει ότι ε, γινόταν κάποια συζήτηση. Βέβαια, πάρα πολύ τιμά ήταν τα σχόλιά σας για την προθεσμία. Οπότε, θα έλεγα, από τη στιγμή που θα είναι διαθέσιμες οι μεταφράσεις, να έχουν οι βουλευτές δύο εβδομάδες κατελάχιστον για να καταθέσουν τροπολογίες. Σε όλες τις γλώσσες νομίζω ότι θα έχουμε τις μεταφράσεις στις 19 Οκτωβρίου. Το αφήνω στη δική σας διακριτική ευχέρεια. Η πράσινη εβδομάδα είναι εργάσιμη, ώστε να έχουμε τουλάχιστον δύο εβδομάδες μετά τις μεταφράσεις. Σας ευχαριστώ για την πρότασή σας. Η κυρία Μέρκης έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον εισηγητή και τους συναδέλφους για την πολύ ωραία συζήτηση. Λίγες παρατηρήσεις. Έχουμε, κατάγομαι από μια όλο και πιο ευρωσκεπτιστική χώρα. Ε, αλήθεια είναι αυτό και ανησυχητικό είναι, τέλος πάντων. Θέλω λοιπόν να πω ότι στηρίζω πάρα πολύ τους στόχους που έχει αναφέρει ο εισηγητής, αλλά συμφωνώ και με όσους συναδέλφους είπαν ότι δεν θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ περιοριστικοί και να υπαγορεύουμε τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να πετύχουμε την ενεργειακή απόδοση. Θα πρέπει δηλαδή να επιτρέψουμε να υπάρχει διαφοροποίηση. Παραδείγματο χάρη στη χώρα μου έχουμε σημαντικά ποσοστά συμπαραγωγής ε, και σε άλλες χώρες. Αφήστε λοιπόν κάποιο περιθώριο ελιγμών για κάθε κράτος μέλος. Θα ήταν σοφό κάτι τέτοιο. Δεύτερον, συλλογική παροχή ισχύω, ε, συλλογική ενεργειακή απόδοση. Ε, συχνά γίνεται λόγος ε, για το συλλογικό επίπεδο, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο και το μικρό επίπεδο. Οι εξοικονομίες ενέργειας, κατά την άποψή μου, δεν γίνονται πάντοτε ε, με δημόσιο τρόπο, συλλογικά, σε μεγάλη κλίμακα. Θα πρέπει να δούμε και το πιο μικρό επίπεδο και να βρούμε και κίνητρα τα οποία θα δώσουμε. Δεν υπάρχει αρκετή αιστεία της πολιτικής μας σε αυτήν την κατεύθυνση. Μία μόνο φορά μπορεί κανείς να δαπανίσει τα χρήματά του. Άρα θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε και την πιο μικρή κλίμακα που μπορούμε εκεί να δώσουμε κίνητρα που θα ήταν ίσω πιο αποδοτικό από του μεγάλου σταθμού. Επίση, ενεργειακή παινία επίση είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Εγώ προέρχομαι, όπω είπα, από ένα κράτο μέλο. Ε, συγκεκριμένο, οι περισσότεροι είναι ενοικιαστέ και όχι ιδιοκτήτε σπιτιών. Και τα πιο πολλά σπίτια είναι παλιά. Αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, ιδίω λόγω τη ε, κατάσταση οικονομική ε, των ανθρώπων οι οποίοι νοικιάζουν η μικροπαραγωγή είναι κάτι σημαντικό. Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με την απόδοση, αλλά και τη δυνατότητα αυτών που νοικιάζουν ένα σπίτι να παράγουν ενέργεια από μόνοι τους. Τελευταίο. Για να εργαστούμε και να συνεργαστούμε καλά, θα ήθελα να συμφωνήσω με την κυρία Φόρτ. Δηλαδή, η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών να μετατεθεί για τις 3 Νοεμβρίου. Αυτό εκ μέρους των σοσιαλιστών. Ευχαριστώ. Ουλτσκοκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι η οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα θα είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αφορά κάτι, κάτι που, μια σειρά μέτρων που μπορεί να οδηγήσει σε συγκεκριμένα σε αυτά αποτελέσματα. Όπως είπαν και, άλλοι βουλευτές, αυτό είναι κάτι το οποίο θα δεσμεύσει και θα εμπλέξει όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε φορά λοιπόν που θα παίρνουν το το λογαριασμό για την κατανάλωση ενέργειας θα έχουν και ένα παραπάνω λόγο να κάνουν κάτι για να αλλάξουν την καθημερινή τους ζωή. Αν πάρουμε λοιπόν αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους να κινηθούν προς την κατεύθυνση αυτή, αυτό μπορεί να είναι πάρα πολύ θετικό και σημαντικό. Τα τελευταία χρόνια έχουμε πει πολλές φορές ότι 1% μικρότερη κατανάλωση ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιστοιχεί σε 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Μπορεί να υπάρχουν και άλλα στοιχεία, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι αρκετά ισχυρό επιχείρημα για να καταδείξει ότι η αποτελεσματικότητα στη χρήση της ενέργειας είναι πολύ σημαντική. Μιλάμε για σημαντικά αποτελέσματα σε εξοικονόμηση χρημάτων, μεγάλη επίπτωση στο περιβάλλον. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, να εξασφαλίσουμε ότι θα κάνουμε τις σωστές κινήσεις. Και εδώ έχουμε λοιπόν στο σχέδιο οδηγίας και στο στόχο αυτής της οδηγίας. Εγώ νομίζω θα ήταν κρίμα αν κάτι τόσο σημαντικό θα το θα μας φέρει σε μια πιο δύσκολη κατάσταση έναντι του Συμβουλίου από ό,τι είμαστε ήδη. Πρέπει να έχουμε σαφείς στόχους για την ενεργειακή απόδοση. Το να μπούμε σε πάρα πολλές λεπτομέρειες μπορεί να πετάξει έξω το βρέφος με τα ύδατα κολύμβησής του. Ξέρω ότι το Σουηδικό Κοινοβούλιο έχει με ευρία πλειοψηφία λάβει αποφάσεις εναντίον ορισμένων στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτή την οδηγία. Δεν ξέρω το σχέδιο οδηγίας, δεν ξέρω αν η Κομισιόν έχει να, να πει κάτι σχετικά. Η δική μου πρόταση βέβαια, η οποία ανα, αντανακλάται και σε αυτά που είπαν άλλοι συνάδελφοι. Είναι ότι η Καλές αποφάσεις πρέπει να έχουν δεσμευτικούς στόχους, αλλά όχι δεσμευτικές λεπτομέρειες, όπως είναι η υποχρεωτική ανακαίνιση 30% των τετραγωνικών των δημοσίων κτίριων. Αυτά δεν είναι πράγματα που πρέπει να τα αποφασίζουμε εμείς. Από την άλλη πλευρά θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε περισσότερο την ιδέα της υποχρέωσης προγραμμάτων για εξοικονόμηση, για μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα. Με την ακρόαση που κάναμε πρόσφατα για την ενεργειακή απόδοση, οι εμπειρογνώμονες οι οποίοι συμμετέσχαν φαίνεται να συμφωνούσαν ε, ότι υπάρχουν σημαντικά πλεονεκτήματα που μπορούμε να αποκομίσουμε από την επιβολή συστημάτων ενεργειακής υποχρέωσης και όλα αυτά δημιουργούν περισσότερες πράσινες θέσεις εργασίας. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να προσθέσει θετικά στοιχεία στην οδηγία για την ενεργειακή απόδοση, το να έχουμε δεσμευτικές ρήτρες χωρίς όμως να έχουμε λεπτομέρειες και υπερβολικές λεπτομέρειες και να υπαγορεύουμε πώς θα γίνουν όλα αυτά. Θέλω να ευχαριστώ τον Κλωτ Τούρμες για το, την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει. Στάθηκε πολύ ανοιχτός προς όλους μας. Όλοι αυτοί που θέλανε να συμμετάσχουν έχουν ήδη συμμετάσχει, έχουν εμπλακεί στην εκπόνηση αυτής της έκθεσης. Πολλοί στους σοσιαλιστές είναι πεπισμένοι ότι πρέπει να είμαστε ηγέτες και πρωτοπόροι στην ενεργειακή απόδοση. Είναι καλό και για τους πολίτες μας και για τη βιομηχανία μας και για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής. Ευχαριστώ. Ο Κλωτούρμες για διαδικαστικό. Πριν έρθουμε στο τέλος της ε, συνεδρίασής μου, θα ήθελα να έχω μια σαφή ε, απόφαση για το πότε θα είναι η προθεσμία τροπολογιών. Έχει προταθεί τώρα μόλις η 3η Νοεμβρίου. Θα ήθελα να ξέρω πότε όμως είναι η οριστική προθεσμία για να μπορέσουμε να αρχίσουμε να εργαζόμαστε και να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Ο κύριος Πίπερ, διαδικαστικά. Έχουμε τρεις συναδέλφους που θέλουν να μιλήσουν επί της ουσίας, δεν βλέπω να προφταίνουν μια συμβαστική πρόταση έχω κάνει, μάλλον την κατάλαβα αυτή, διαφορετικά την πρόταση αυτή, δύο εβδομάδες μετά από τη στιγμή που θα είναι διαθέσιμες οι μεταφράσεις. Αυτή ήταν η συμβιβαστική λύση που, που, προτάθηκε, αλλά υπάρχουν και άλλες προτάσεις που έχουν γίνει, από ό,τι ξέρω, λέει και ο Σπίπερ. Υπάρχουν διαφορετικές ε, ερμηνείες. Κυρία διαφόρτη είπε, δύο εβδομάδες μετά την ημέρα που θα είναι διαθέσιμες οι μεταφράσεις. Υπήρχε τώρα ο κύριος Τούρμες χωρίς μικρόφωνο. Χωρίς μικρόφωνο. Για τις 19 θα είναι διαθέσιμες οι μεταφράσεις για όλες τις γλώσσες. Οπότε ερχόμαστε στις 3 ή στις 4 Νοεμβρίου. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Θα πρέπει να σταματήσουμε όλες αυτές οι οικοτολογίες σε σχέση με τις προθεσμίες. Η, το παιχνίδι αυτό με τις προθεσμίες ξεκινά από σένα, γιατί εσύ έθεσες κάποιες προθεσμίες χωρίς να συζητήσεις με κανένα, ούτε με μένα. Όλα είχαν προετοιμαστεί και πριν από την μια εβδομάδα την προηγούμενη Παρασκευή είδα ότι δεν υπάρχει η έκθεση. Και είπα στη γραμματεία μπορώ να την αφήσω στην ημερησία διάταξη τη στιγμή που δεν υπάρχει έκθεση ακόμα έτοιμη. Παρ' όλα αυτά έκανα σήμερα τη συζήτηση. Παρά το γεγονό ότι δεν υπήρχε έκθεση. Αυτό είναι το πρώτο. Μιλάω για τα γεγονότα. Να είμαστε σαφεί. Κανονικά η διαδικασία προβλέπει ότι όλοι οι συνάδελφοι θα πρέπει να έχουν την έκθεση στην δική τους γλώσσα προτού ξεκινήσουν οι συζητήσεις. Αν λοιπόν στις 19 του μηνός έχουμε όλα τα κείμενα στις γλώσσες των βουλευτών, αν έχετε στις 20 όλη την έκθεση, μπορούμε να κάνουμε για πρώτη φορά την λεπτομεριακή συζήτηση για την έκθεση αυτή. Αυτό είναι σωστό. Και τότε μπορείτε να αποφασίσετε αν θα δώσετε μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες, πόσο καιρό χρειάζεται κανείς για να διατυπώσει τις τροπολογίες του. Και εδώ βλέπω ότι υπάρχει ποικιλία απόψεων. Υπάρχει μια... Δεν υπάρχει ομοφωνία. Άλλοι λένε ότι δεν χρειαζόμαστε χρόνο, άλλοι λένε χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το θέμα αυτό και όλα αυτά πρέπει κάπως να τα συγκεράσουμε, να καταλήξουμε σε κάποια λύση. Υπάρχουν ε, οι δυνατότητες μιας ε, συνένεσης ή αν δεν έχουμε συνένεση πρέπει να ψηφίσουμε και να αποφασίσουμε. Πάλι διαδικαστική παρέμβαση. Η κυρία Χολ πρώτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκτιμώ όλους ιδιαίτερο την προθυμία των συναδέλφων από όλε τι πλευρέ ε, να συζητήσουμε το θέμα επικοδομητικά. Για να ε, διευκολύνουμε την όλη συζήτηση, καλό θα ήταν πράγματι να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. ακούγοντα. τι είπε η συνάδελφο Βίκυ Φόρτ και η Γιούντιτ Μέρκη, ουσιαστικά για το ίδιο μιλάμε όλοι. Δηλαδή θέλουμε ε, να έχουμε μετά την ημερομηνία που θα έχουμε τις μεταφράσεις 19 Οκτωβρίου, δύο εβδομάδες στη θέση μας, άρα 3 Νοεμβρίου για τις τροπολογίες. Το μόνο που σας ζητάω, κύριε Πρόεδρε, είναι να το πείτε έτσι ξεκάθαρα, έξω από τα δόντια. Πρέπει ε, να έχουμε ε, ημερομηνίες. Γιατί έχουμε δύσκολο πρόγραμμα, είναι φορτωμένη η ατζέντα μας. Πρέπει να ξέρουμε πότε έχουμε τι. Γιατί τελικά μου φαίνεται ότι ενώ μιλάμε όλοι για το ίδιο πράγμα, ε, δεν μας έχετε διευκρινίσει. Καλό θα ήταν να μας πείτε. 3 Νοεμβρίου, δηλαδή έχουμε δύο εβδομάδες μετά τις μεταφράσεις, για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Κυρία Μέρκης, ευχαριστώ πρόεδρε. <clears throat> Υποστηρίζω αυτή την πρόταση. Δεν νομίζω ότι υπήρξε κάποια παρανόηση. Υποστηρίζω την κυρία Χολ και την κυρία Φόρτ. 3 Νοεμβρίου λοιπόν. Και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι Πρόκειται για το δύο εβδομάδες μετά τη διαθεσιμότητα των μεταφράσεων και όλοι θα θέλαμε πράγματι να έχουμε σαφήνεια και οριστικότητα για την ημερομηνία αυτή. κυρία Κολάσκα Μπομπίνσκα. Κοιτάξτε, αυτό είναι πολύ κακό για την έκθεση και για ένα ε, θέμα που τελικά αντί να το συζητάμε, συζητάμε όλο τις ημερομηνίες πριν, μετά γιατί δεν μπορούμε να τηρήσουμε την κανονική διαδικασία και έτσι προσπαθούμε να πιέσουμε προς μια κατεύθυνση και υπάρχει κάποιος εκνευρισμός. Εγώ θα έλεγα όσοι οι ομιλητές δεν έλαβαν το λόγο να μπορούσαμε να λάβουμε το λόγο στη συζήτηση. Αλλά σε ό,τι αφορά τις προθεσμίες είπαν κάποιοι ότι είναι μια εβδομάδα πράσινη μέσα σε αυτή την προθεσμία. Θα πρέπει να αποφασίσουμε. Εδώ πέρα καθόμαστε... Ε, ή πάμε στην ε, περιφέρειά μας και μιλάμε με τους ψηφοφόρους μας ή καθόμαστε εδώ και κάνουμε τροπολογίες. Λοιπόν, εγώ δεν ε, θέλω αυτή την πολύ σημαντική δουλειά να την επιταχύνουμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές οικονομικές επιπτώσεις, υπάρχουν επιπτώσεις του πολίτε για την αυτοδιοίκηση, τη διαχείριση. Ευχαριστώ. Για να μην κρατήσει για πολλή ώρα αυτό το πράγμα, επανέρχομαι σε αυτό που είπε η κυρία Φορ. Θέλω όλοι να έχουν τα ίδια δικαιώματα, όλα τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν και εγώ ενοχλήθηκα τις τελευταίες μέρες γιατί είχαμε πάρα πολλά email, πάρα πολλές παρεμβάσεις για την ημέρα διάταξη. Δεν μου φάνηκε αυτό διασκεδαστικό. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει μια ανάγκη να περιμένουμε δύο εβδομάδες μετά από την μετάφραση των κειμένων. Όλοι ξεκινάμε με την υπόθεση ότι θα έχουμε 19, του μηνός θα έχουμε την ε, μετάφραση. Αυτό μας οδηγεί στις 3 Νοεμβρίου. Είπε η κυρία Κολάσκα, Πομπίνσκα, ότι υπάρχει το θέμα της πράσινης εβδομάδας. Μπορούμε να βρούμε μια λύση για το θέμα αυτό. Έχω την εξή ιδέα. Να πούμε 19 Οκτωβρίου συν δύο εβδομάδες και να περάσουμε στην Δευτέρα, γιατί όλοι οι συνάδελφοι μπορούν να είναι εδώ τη Δευτέρα και να υπογράψουν. Δύο μέρες. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα για δύο μέρες. Γιατί έτσι δεν έχουμε και το πρόβλημα με την πράσινη εβδομάδα. Ο Κλωτούρμες δεν συμφωνεί μάλλον. Δεν θέλω να τρομοκρατήσω κανένα ή να επιβάλλω κάτι. Αν καθυστερήσουμε ακόμα, δεν θα είμαστε έτοιμοι εγκαίρως. Εγώ νομίζω ότι τώρα θα πρέπει να αποφασίσουμε και αν δεν υπάρχει συνένεση να ψηφίσουμε. Εντάξει, αυτό περίμενα κι εγώ. Ο κύριος Πίπερ. Ποιος έχει καθυστερήσει τρεις εβδομάδες για την έκθεση. Γιατί βρισκόμαστε εδώ. Εσείς έχετε προκαλέσει την καθυστέρηση τριών εβδομάδων. Και τώρα δεν μας δίνεται τη δυνατότητα να έχουμε δύο εβδομάδες για να κοιτάξουμε την έκθεση. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Ε, στείλαμε 16 με 18 ερωτήσεις στην Κομισιόν για τα θέματα αυτά και δεν πήραμε απαντήσεις. Θα ήταν χρήσιμο να έχουμε τις απαντήσεις. Θα ήταν απλώς μια ιδέα. Πάρα πολλοί ζητούν το χρόνο. Λοιπόν, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Ξαναλέω ποια είναι η πρότασή μου. μπορούμε να συμφωνήσουμε μετά τη μετάφραση 19 Οκτωβρίου δύο εβδομάδες και περνάμε στην επόμενη Δευτέρα ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα με την ε, πράσινη εβδομάδα. Για να μην μπορεί να πει κανείς ότι δεν μπορεί να είναι εδώ την εβδομάδα αυτή να, ε, να υποβάλει την πρόταση αυτή, να υποβάλει τις τροπολογίες μέχρι την επόμενη Δευτέρα. Υπάρχει κανείς κατά αυτής της λύσης. Δευτέρα μετά στις 7. 7 του μηνός. 7 του μηνός. 7 Νοεμβρίου. 12 η ώρα το μεσημέρι τη Δευτέρα, 7. Μπορούμε να συμφωνήσουμε, ο Κλοντ. Εγώ συμφωνώ μόνο με την προϋπόθεση ότι θα ψηφίσουμε το αργότερο τον Ιανουάριο. Γιατί πρέπει να σταματήσουμε αυτό το παιχνίδι. Εάν πούμε 7 Νοεμβρίου θα πει αυτό ότι το αργότερο θα ψηφίσουμε το Γενάρη. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια συμβιβαστική πρόταση. Ο πρόεδρος, δεν ξέρω πότε θα τελειώσουμε αυτό το παιχνίδι. Κάποιοι παίζουν παιχνιδάκια εδώ πέρα. έχω κάποιες ε, δικές μου ιδέες, αλλά τις βάζω κατά μέρος. Αν υποθέσουμε ότι όλοι είμαστε σοβαροί, και φυσικά θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να ολοκληρώσουμε για να μπορέσουμε τα αποτελέσματα αυτά να τα χρησιμοποιήσουμε στην, επόμενη Προεδρία. Επιμένει, πρέπει να λυθεί το θέμα επιδανική Προεδρίας και αν έχω καταλάβει καλά δεν είναι και κανείς αντίθετος με αυτή την ιδέα όσο το νωρίτερο τόσο το καλύτερο. Από ό,τι κατάλαβα όμως υπάρχουν θέματα και θέματα ουσία τα οποία τίθενται και ο ίδιος ο ορισμός της ενεργειακής απόδοσης τίθεται και θα πρέπει να συζητήσουμε και με τους εμπειρογνώμονες. Λοιπόν, ξαναρωτάω, συμφωνείτε, συμφωνείτε να επιλέξουμε την προθεσμία 7 Νοεμβρίου 12 το μεσημέρι για τις τροπολογίες. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Έχουμε δύο-τρία λεπτά ακόμα μετάφρασης. Παρακαλώ, οι υπόλοιπε ε, παρεμβάσεις να γίνουν κάποια άλλη στιγμή και να σας υπενθυμίσω το ψήφισμα για τη COP17 να θεωρήσουμε ότι το έχουμε εγκρίνει. Ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους που δεν μπόρεσαν να λάβουν το λόγο. Εντάξει, ελπίζω ότι η γραμματεία έχει καταγράψει τα ονόματά σας να μπορέσετε να μιλήσετε την άλλη φορά. Αλλά πρέπει να είστε παρόντες βέβαια στην επόμενη συζήτηση.